Από ό,τι καταλαβαίνω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σίγουρα θα έρθουν και κάποιοι συνάδελφοι. Είναι στο δρόμο τους από την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά δεν έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε αμέσως την ε, συνεδρίαση. Θα θυμάστε ότι πριν το διάλειμμα είχα ξεκινήσει να παρουσιάζω το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, τις ανακοινώσεις μου, θα ήθελα να τις περατώσω να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από τους συντονιστές κατά τη συνεδρίαση που είχαμε χθες το βράδυ. Ήδη σας είπα τι θα γίνει με το Ταμείο Αλληλεγγύης το πρωί. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι επίσης συζητήσαμε τις μη νομοθετικές γνωμοδοτήσεις και οι συντονιστές αποφάσισαν ότι σχέδια γνωμοδοτήσεων και εκθέσεις ιδέας πρωτοβουλίας από άλλες επιτροπές όπως περιβάλλοντος δημόσιας υγείας, ασφάλεια τροφίμων ή με βάση τη λευκή βίβλο της ε, Επιτροπής για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Όλα αυτά είναι θέματα που θα τα αναλάβουν ε, οι σοσιαλιστές. Επίσης, συμφωνήσαμε στη συνεδρία των συντονιστών ότι η έκθεση για την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κοινοτική προσέγγιση για τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μάλλον θα αναλυθεί από την ομάδα των φιλελευθέρων. Όμως αυτό έχει να κάνει και με μια άλλη γνωμοδότηση, όπου και πάλι υπάρχει μια προτίμηση για την άλλη. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και στις δύο περιπτώσεις, τι θα αποφασίσει και η ίδια η ομάδα των φιλελευθέρων για το ποια γνωμοδότηση θα αναλάβει. Πιστεύουμε όμως ότι και τις δύο η Άλντε θα τις πάρει. Επίσης με την Επιτροπή της Γεωργίας έχουμε μια γνωμοδότηση. Γεωργία σε περιοχές με φυσικές με φυσικά μειονεκτήματα. Εδώ θα αναλάβει το ΕΛΚ και μια τέταρτη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και το βιώσιμο, μάλλον το βιώσιμο μέλλον των μεταφορών είναι το θέμα της. Δεν είναι απόλυτο σαφέ ακόμη. Ποιο αναλαμβάνει, υπάρχουν πολλέ πολιτικέ ομάδε που τη θέλουν. Θα σα ενημερώσω λοιπόν αργότερα, μόλι ληφθεί τελική απόφαση, για το ποια πολιτική ομάδα θα αναλάβει αυτήν την ε, έκθεση. Τώρα, για τι εκθέσει πρωτοβουλία οι συντονιστές συμφώνησαν για μια σειρά προτάσεων και λήφθη απόφαση για εκθέσει ιδίας πρωτοβουλία που θα αναλάβει το ΕΛΚ καταρχάς. Έκθεση για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να αντιμετωπίσουμε την τωρινή κρίση και τις διαφορετικέ προσαρμογές που θα χρειαστούν την εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προποθέσει για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα σε διεθνή κλίμακα και τις εκθέσει υλοποίησης. Το ΕΛΚ λοιπόν θα έχει δύο εκθέσει πρωτοβουλίας, καθώς και μια έκθεση υλοποίησης για το συντονισμό μεταξύ του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Οι Σοσιαλδημοκράτε έχουν προτείνει δύο εκθέσει για του στόχου τη Λισαβόνα η μία και η άλλη για την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή τη Βαλτική θάλασσας. Η Άλντε ακόμη έχει, είναι διχασμένη μεταξύ δύο εκθέσεων, είτε τη στρατηγική για την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών ή την καλή διακυβέρνηση σε σχέση με την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. Στη γραμματεία περιμένουμε την απόφαση των συναδέλφων για το ποια τελικά θα αναλάβουν, ποια θα συντάξουν. Η πράσινη διαφάνεια για την περιφερειακή πολιτική και τη χρηματοδότησή της. Οι συντονιστές αποφάσισαν να, συναντήσουν, να συζητήσουν ε, μελλοντικά μία ακόμη έκθεση που πρότειναν οι πράσινοι για τους νέους δείκτες για τη μέτρηση των κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των περιφερειών και για το μέλλον. συμφωνήσαμε ότι όσο το δυνατόν συντομότερα οι ομάδες θα στείλουν τις προτάσεις τους για το 2010 οι οποίες θα πρέπει να σταλούν πριν την συνάντηση του Νοεμβρίου της Επιτροπής Περιφερειών, της Επιτροπής Ρέτζη μάλλον, και όλες οι ιδέες για εκθέσεις νομοτήσεις πρέπει να έχουν φτάσει στο Νοέμβριο. Αν δεν υπάρχει λοιπόν αντίρρηση, οι συντονιστές, οι αποφάσεις μάλλον των συντονιστών θεωρούνται εγκεκριμένες και θα περιμένουμε απλώς τις τελικές αποφάσεις κάποιων συναδέλφων όταν θα είναι έτοιμοι. Το σημείο λοιπόν αυτό της ημερήσιας διάταξης το έχουμε ολοκληρώσει, περνάμε στο 5. Η μειωμένο συντηλεστή ειδικού φόρου κατανάλωση στη Μαδέρα. Έχουμε μαζί μα τον κύριο Έλλη Ωράου, ο συγκεκριτής είπε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων σήμερα. Είναι μια πρόταση χωρί πολλέ που δεν είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη. Το ΕΛΚ πρότεινε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό ε, στα πλαίσια της απλουστευμένης διαδικασίας χωρίς τροπολογίες. Και εάν συμφωνείτε, αυτό και θα κάνουμε. Να ρωτήσω τον κύριο Έλλη Ορό εάν θέλει να σχολιάσει. Ναι, Πρόεδρε. Συμφωνώ με την απλουστευμένη διαδικασία και την επιλογή αυτή. Λίγα λόγια ίσως για να παρουσιάσω την έκθεση να πω ότι η παραγωγή είναι ο πνευματοδόν και ειδικό ρουμνιού είναι σημαντικό όχι μόνο για τις ε, Ασόρες και τη Μαδέρα, αλλά και στις Αντίλες και στο νησί της Ρεουνιών. Πιστεύουμε ότι το προτινόμενο μέτρο θα πρέπει να ανασταλεί, να καταργηθεί μάλλον, ώστε ο τομέας αυτός να διατηρήσει την ποιοτική του παραγωγή, αλλά και να διαφυλάξουμε ένα μέσο το οποίο επιτρέπει να αντισταθμίσουμε τις υψηλότερες τιμές των ε, ενοπνευματοδών αυτών που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό και μετά από συζητήσεις και διαβουλεύσεις με συναδέλφους Πορτογάλους από τη Μαδέρα και τις Ασόρες αποφασίσαμε να έχουμε αυτή την επιτεχημένη διαδικασία, την απλουστευμένη διαδικασία Κάτι το οποίο μας βρίσκει απολύτω σύμφωνος. Για όλους αυτούς τους λόγους θα κατανοείτε αγαπητοί συνάδελφοι ότι σας ζητώ να στηρίξετε αυτήν την έκθεση. Ιδού. Τώρα, εάν οι συνάδελφοι από τις συγκεκριμένε περιοχές θέλουν να λάβουν θέση, φαντάζομαι ότι η άποψή τους είναι ενδιαφέρουσα για όλους. Αυτά ήθελα να πω, Πρόεδρε, εντάχει. Κύριε Τεσέιρα. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να χαιρετήσω τον κύριο Όραο, με τον οποίο συνεργάστηκα για την επεξεργασία του θέματος και τον ευχαριστώ για την προσοχή και το ενδιαφέρον που έδειξε για την προετοιμασία αυτή. Να σας πω τα εξής πολύ σύντομα. Η πρόταση αυτή έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις για την περιοχή της Μαδέρας και των Ασορών. Στην Πορτογαλία επήγει να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή. Θέλουμε λοιπόν ο μειωμένος συντελεστής να ισχύσει κάτι που είχε ξεκινήσει να ισχύει από το 2002. Στην Πορτογαλία η κατανάλωση των προϊόντων αυτών που έχουν παραχθεί στη Μαδέρα και τις Ασόρες υπόκειται σε ειδικό καθεστώς. Η, με, το, με τον κανονισμό 81-2008 έληξε η ισχύ του καθεστώτος αυτού. Τώρα θέλαμε λοιπόν να προβλέψουμε το 2009 με ένα δρομικό ε, με αναδρομική ισχύ την ε, υλοποίηση του κανονισμού του 2003 ξανά. Έτσι λοιπόν με την κατάργηση αυτή τα πλεονεκτήματα του 2002 θα διατηρηθούν και θα σεβαστούμε τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητε των, ε, των απομακρυσμένων αυτών περιοχών, οι οποίες έχουν ε, την ιδιαιτερότητα να παράγουν τα προϊόντα αυτά σε μικρέ εκμεταλλεύσει, πολύ μικρές επιφάνειες. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά έλαβε υπόψη τι ιδιαίτερότητε τη παραγωγή των προϊόντων αυτών στα αρχιπελάγη και εδώ δεν νομίζω ότι έχουμε καμία περίπτωση αθέμη ανταγωνισμού, καμία δυνατότητα ανάπτυξη τέτοιου ανταγωνισμού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν πώ θα διαμορφωθεί το καθεστώ πώληση των προϊόντων αυτών, γιατί θα καθορίζει την παραγωγικότητα των νήσων αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι όπω προτείνει ο εισηγητή, ο κύριο Οράου, η νέα πρόταση δεν απαιτεί καμία τροποποίηση και απλώς θα ήθελα να ζητήσω την στήριξη των συναδέλφων να παραμένουν στο άρθρο 48 του κανονισμού και στην αποστευμένη διαδικασία. Εάν συμφωνείτε λοιπόν, Πρόεδρε, θα θέλαμε η πρόταση αυτή να εγκριθεί χωρίς τροποποίησης. Και η έκθεση αυτή να υποβληθεί στην Ολομέλεια ή δυνατόν ήδη τον Οκτώβριο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Μπορούμε λοιπόν να ομόφωνα να αποδεχτούμε αυτή την απόφαση και να στείλουμε την πρόταση στην Ολομέλεια. Πρόεδρε, να προσυπογράψω και εγώ εξ ονόματος των σοσιαλιστών, των σοσιαλδημοκρατών, στην απλουστευμένη διαδικασία και την επιλογή της. Γιατί το προϊόν αυτό είναι, είναι σημαντικό για τη Μαδέρα, υπήρχε ήδη καθυστέρηση και υπάρχει σοβαρό αντίκτυπο στι μικρέ τοπικέ κοινωνίε. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα. Θέλουμε λοιπόν η έκθεση να μείνει ω έχει και ζητούμε τη στήριξη για την έγκριση. Και τώρα, άλλο κανεί άλλος κανείς που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ωραία, λοιπόν, ομόφωνα εγκρίνουμε την απόφαση, τη στέλνουμε στην Ολομέλεια και σα ευχαριστώ. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στο σημείο 12. Εάν ε, είναι μαζί μα, ο Καρή Μαντέλη η Μαντέλη. Εδώ είπαμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή και του εισηγητή, αν και αυτή την έκθεση τη δούμε τον Νοέμβριο και θα την ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Όμω σήμερα θα ήθελα να ανοίξω τη συζήτηση και να ζητήσω από την κυρία Ντελή να μα παρουσιάσει το σημείο αυτό. Ναι, θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το 2011 να κηρυχθεί το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Η πρόταση απόφαση της Επιτροπής είναι συνέχεια μιας κήρυξης του Κοινοβουλίου της Δευτέρας ε, Σεπτεμβρίου 2008 ώστε να κηρυχθεί το έτος 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις ανταλλαγές εμπειριών, καλών πρακτικών και τις ε, προσπάθειες προς μίμηση από τα κράτη-μέλη για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές αλλά και την κοινωνία των πολιτών ώστε να δημιουργηθούν οι πρόσφορες συνθήκες για τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή θέλει με τον εθελοντισμό να εκφραστεί ενεργά η συμμετοχή των πολιτών η οποία θα εδραιώσει τις κοινέ αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εθελοντισμός λοιπόν θα επιτρέψει να ενθαρρύνουμε τις θεμελιώδεις αξίες όπως ε, η ιδιότητα του πολίτη, η αλληλεγγύη, η υπεράσπιση του κοινού συμφέροντο και η μη διάκριση. Είναι σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη και άλλα σκέλη όπω η εκπαίδευση, η παιδεία, το περιβάλλον, η υγεία, ε, η πολιτική ανάπτυξη, η ισότητα ευκαιριών, οι εξωτερικέ σχέσει. Ο εθελοντισμό μπορεί επίση να ε, συμβάλλει στην αρμονική ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Τέσσερις είναι οι στόχοι οι οποίοι προτείνονται από την Επιτροπή σε αυτήν την πρόταση απόφασης. Καταρχάς, να εργαστούμε ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο που θα ευνοήσει την δημιουργία του εθελοντισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, να προσφέρουμε στι οργανώσει εθελοντών τα μέσα για να εργαστούν και να βελτιώσουμε την ποιότητα του εθελοντισμού. Έπειτα, να εξισορροπήσουμε τι δράσει του εθελοντισμού, να τι ανταμείψουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για την προστιθέμενη αξία και την εμβέλεια του εθελοντισμού. Έτσι λοιπόν, συγκεκριμένε δράσει μπορούν να αναλυφθούν ώστε να επιδιώξουμε του στόχου αυτού, όπω πρωτοβουλίε διοργανωμένε σε όλα τα επίπεδα, διοικητικό, κοινοτικό δημοτικό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011 θα πρικοδοτηθεί από έναν προπολογισμό 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή προτείνει εδώ να προσταθούν 2 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών εργασιών και βάση του προσχεδίου προπολογισμού του 2010. Όλοι αυτοί οι στόχοι είναι ευγενείς και ο φιλαντισμό θα είναι ένα καθοριστικό εργαλείο για να προωθήσουμε την κοινωνική συνοχή μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών για την ε, εκπαίδευση των πολιτών και για όλους τους μη κερδοσκοπικούς ε, στόχους που είναι τόσο αναγκαίοι και λείπουν στους καιρούς μας. Πέρα λοιπόν από το θέμα των μέσων και τον προπολογισμό των 6 εκατομμυρίων ευρώ, Φαίνεται ανεπαρκέ κάτι τέτοιο σε σχέση με τι προκλήσει του εθελοντισμού. Ένα τέτοιο ευρωπαϊκό έτο θα πρέπει να είναι ευκαιρία για να βεβαιώσουμε και να επανεπιβεβαιώσουμε κάποιε καθοριστικέ αρχέ και αξίε, οι οποίε δεν διακριβώνονται επαρκώ στο κείμενο που μα έχει προτείνει η Κομισιόν. Ε, εδώ πρέπει να καταλάβουμε καλά τι εννοούμε με τον εθελοντισμό. Θα πρέπει λοιπόν εκ των προτέρων να αποσαφηνίσουμε το, νομικό καθεστώς του εθελοντισμού. Διακρίνουμε τι είναι εθελοντισμός και να μην επιτρέψουμε δύο αυτές έννοιες να, να υποκαταστήσουν τις αμοιβόμενες υπηρεσίες ή τις κοινωνικές υπηρεσίες ή την ε, δημόσια δράση. Ο εθελοντισμός υπό την έννοια της πρότασης της Επιτροπής πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις δύο έννοιες. Έπειτα ένα σημείο πρωταρχική σημασία. Το Ευρωπαϊκό Έτο Εθελοντισμού θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για να εγγυηθούμε την προστασία των καταναλωτών ε, ω προ την εργασιακή ασφάλεια, την υγεία και την κοινωνική προστασία. Εάν είναι υπέρμετρο ο αριθμό των εθελοντών, υπάρχει περίπτωση ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των αποστολών που αναλαμβάνουν και δεν θα υπάρχει και εγγύηση ή κάλυψη για αυτού. Επίση, ο εθελοντισμό θα πρέπει να μπορεί να ε, συμπεριληφθεί σε ένα σχέδιο διαδικασιών και μάλιστα σε ένα ολόκληρο πρόγραμμα ζωή. Γι' αυτό θα πρέπει κανεί να διευκολύνει την αναγνώριση του εθελοντισμού, την ε, αξιοποίηση και την αναγνώριση των αξιών και να αναζητήσει ισοδύναμα κατά τη διάρκεια των μαθησιακών κύκλων που να καταλήγουν σε επαγγελματικέ διεξόδου. Επίση, κάτι άλλο που θα είναι εύστοχο είναι να διευκολύνουμε την πρόσβαση των οργανώσεων εθελοντών σε χρηματοδοτήσει επαρκή και αηφόρου, χωρί να του επιβάλλουμε πολύ επαχθεί διοικητικέ διαδικασίε και με όλου του απαραίτητου ελέγχου για τι δαπάνε εννοείται των δημόσιων κοντιλίων. Επίση, πρέπει να καταπολεμήσουμε όλε τι μορφέ διάκριση κάποια κρατημέλη απαγορεύουν την άσκηση του εθελοντισμού στους ε, αλλοδαπούς κατοίκους. Οι υπηρεσίες των Ευρωπαίων Εθελοντών ε, αποκλείουν λόγω χάρη τους επικούς ε, τρίτων κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2011 θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για να αναμονήσουμε αυτές τις πρακτικές και να επιτρέψουμε σε κάθε κάτοικο κράτους μέλους, όποια και είναι η εθνικότητά του, το κοινωνικό του καθεστώς, το διοικητικό του καθεστώς, να μπορεί να εξασκήσει άνετα τις εθελοντικέ του διαθέσεις. Μάλιστα, για τον μη κερδοσκοπικό τομέα, ο εθελοντισμό θα πρέπει να επιτρέψει να προωθήσουμε ιδέε και πρακτικέ, οι οποίε είναι απολύτω αναγκαίε στην εποχή μα, όπω η πρόθεση τη ειρήνη, η συνεργασία βορρά και νότου, η προστασία του περιβάλλοντο, ή ακόμη η ανάπτυξη και η αναγνώριση τη κοινωνική οικονομία και τη αλληλεγγύη. Όλε αυτέ οι καθοριστικέ σημασία έννοιε πρέπει να αναφέρονται ρητό στο κείμενο. Το Ευρωπαϊκό Έτο Εθελοντισμού θα πρέπει επίση να διεξαχθεί σε μια διαρκή εταιρική σχέση με τις οργανώσεις των εθελοντών. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε την, ένα ε, σταθερό θεσμικό πλαίσιο για τη συμμετοχή των οργανώσεων αυτό στην δημόσιες διαβουλεύσεις. Ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως την προστιθέμενη αξία του εθελοντισμού θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και μια ειδική κατηγορία στις ε, στατιστικές, στους στατιστικούς υπολογισμούς της Eurostat, ώστε να προβλέψουμε τη συνεισφορά των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, να καλύψουμε τους διάφορους λογαριασμούς των κρατών και το έργο των εθελοντών. Και τα κράτη-μέλη να μπορούν να λάβουν υπόψη την εργασία των μη κερδοσκοπικών οργανισμών στη σχεδιασμό των πολιτικών τους. Τέλος, για να επιδιώξουμε καλύτερα αυτούς τους στόχους, καλό θα ήταν με ευκαιρία του έτους αυτού να προωθήσουμε και την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τους εθελοντές. Κάτι που θα στηρίξει ακόμη περισσότερο το έργο των εθελοντών και τις ευθύνες τους. Βεβαίως, δεν θα αρκέσει ένα και μόνο έτος. Θα πρέπει να καθορίσουμε κοινού στόχους για τις δραστηριότητες των εθελοντών. Πέραν του 2011. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε και να υλοποιήσουμε την ημερομηνία της 5ης Δεκεμβρίου ως ε, μέρα παγκόσμια που από το 85 έχει εγκρίνει ο ΙΕΟΣ μέρα εθελοντισμού. Ε, επειδή μάλιστα ο, χώρος, ο κόσμος της εργασίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος ε, τη σημερινή εποχή. 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε θεωρούνται φτωχοί αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ελληνική μεταξύ γενεών, κοινωνικών τάξεων και εργασιακών δυνάμεων. Θα πρέπει λοιπόν ο εθελοντισμό να χρησιμοποιηθεί ω αφορμή για να ενισχύσουμε του κοινωνικού δεσμού. Όμω δεν μπορεί να είναι το α και το ω μια πολιτική καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις αμοιβόμενες εργασίες και να επιτρέψει στους εργοδότες να έχουν φτηνή και χειραγωγήσιμη εργατική δύναμη στα χέρια τους. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι το 2011 που θα ακολουθήσει το 2010 το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της ένδυας θα εμπίπτει στο σωστό πνεύμα. Πρέπει επίσης να προσδιορίσω ότι ο αριθμός των εισηγητών ε, Επιτροπή Πολιτισμού που ονομάστηκε χθε, ο κύριος Μάρκος Κούρια, μέλος του ΕΛΚ, είναι συγκεκριτής επί της ουσίας, οπότε καθήλων αρμόδιος και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που θα μπορέσω να μοιραστώ την έκθεση αυτή μαζί σας. Ελπίζω, ελπίζω ότι κι εσείς θα με πλουτίσετε με τις προτάσεις σας και ελπίζω να έχουμε μια άριστη συνεργασία σας. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τρεις ευρωβουλευτές ζήτησαν το λόγο. Μην ξεχνάτε ότι εκτενή συζήτηση για το θέμα αυτό θα γίνει το Νοέμβριο, όταν υποβληθεί επίσημα το έγγραφο της γνωμοδότησης. Σας θέρμα παρακαλώ λοιπόν, σήμερα περιοριστείτε σε συγκεκριμένες προτάσεις προς την εισηγήτρια, την κυρία Καρή Μαντελή, ώστε να μπορέσει να τις λάβει υπόψη. Δεν χρειάζεται να χάνουμε το χρόνο μας σε μακροσκελείς δηλώσεις, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ο κύριος Καρόνα. Ε, πολύ σύντομα θα επωφεληθώ τη συζήτηση επί της ουσίας που θα ακολουθήσει. Απλώς να πω σήμερα ότι η συνάδελφος Ντελή με τρόπο πολύ σαφή και πιστικό με τρόπο λοιπόν ε, σαφή και πιστικό παρουσίασε το θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και το γεγονός ότι το 2011 θα έχουμε μια σημαντική ευκαιρία για να δώσουμε την αξία που τους αρμόζει στην ε, εργασία των εθελοντών. Κάτι που πολλές φορές ε, πηγαίνει χαμένο το έργο των εθελοντών. Από αυτή την άποψη λοιπόν αυτή η γνωδότηση είναι χρήσιμη και χρήσιμο θα είναι και η Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως, η δική μας Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως το έτος αυτό έτος, το οποίο πρόκειται να προβλεφθεί. Είναι λοιπόν σημαντικό να αξιολογήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή εάν οι πόροι οι οποίοι έχουν ως τώρα προβλεφθεί, αν είναι επαρκής για να επιδιώξουμε τους στόχους που ε, λεπτομερώς μας κατέδειξε η συνάδελφος. Ε, θα τοποθετηθώ εκ νέου όταν γίνει επί της ουσίας συζήτηση με ενδεχομένως πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, Θα είμαι και εγώ λακωνικός. Καταρχήν, επιδοκιμάζω και επικροτώ αυτή την πρωτοβουλία της Επιτροπής και να επενέσω και την κυρία Χάρκιν που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πρόταση για την ανακήρυξη του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού. Είναι αξιέπινη πραγματικά αυτή η στόχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μακάρι να το υλοποιήσουμε, γιατί κάτι τέτοιο θα σημαίνει αισθητή πρόοδο για το 2011. Μπορεί ο θελοντισμός όχι μόνο να βοηθήσει την οικονομία, αλλά να επισπεύσει και την ανάκαμψη. Και έχουμε την, ε, μία έρευνα από ένα ερευνητικό κέντρο με θέμα τον εθελοντισμό. Και είπε ότι αν εξασφαλίσουμε τον ελάχιστο μισμό, ε, μισθό σε όλους τους εθελοντές ε, θα βελτιωθεί η κατάσταση πάρα πολύ. Και 3 στους 10 Ευρωπαίους είναι εθελοντές. Ενώ 7 με 8 στους 10 έχουν δηλώσει επιθυμία να γίνουν εθελοντές. Αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το 2011, να γεφυρώσουμε το κενό από τους πραγματικούς εθελοντές ε, προς τους επίδοξους εθελοντές και να διευκολύνουμε όσους έχουν αυτή την επιθυμία να την πραγματοποιήσουν. Είναι μοναδική ευκαιρία που έχουμε. Θα πρέπει καταρχήν να αναγνωρίσουμε τον εθελοντισμό, να φέρουμε τον εθελοντισμό κοντά στους πολίτες, ε, να το κάνουμε προσιτό στους πολίτες και να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο όλων των Ευρωπαίων. Τεράστια ευκαιρία λοιπόν μας δίνεται. Θέλουμε να αναμειχθούμε στη διαδικασία αυτή και να την ε, μετατρέψουμε σε εντυπωσιακή επιτυχία για το 2011. κυρία Κάθριν Μπέργκερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να υποστηρίξω τις προσπάθειες αύξησης του προϋπολογισμού για τον εθελοντισμό. Γιατί ε, είναι ποικίλα τα χαρακτηριστικά του κλάδου και καλό θα ήταν να εφοδιάσουμε την πρωτοβουλία αυτή με επαρκή κονδύλια για να αφυπνίσουμε τους Ευρωπαίους ε, ως προς την ανάγκη του εθελοντισμού. Η έκθεση για το ευρωπαϊκό έτος ε, της, ε, του εθελοντισμού με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας θα εμπίπτει στη διαδικασία συναπόφαση και όχι πια της διαβούλευσης. Οπότε η Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να περιμένει ίσως μετά τον Ιανουάριο που θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη πριν οριστικοποιήσει την έκθεσή της έχει περαιτέρω πληροφορίες για αυτό το θέμα, για το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης της Επιτροπής Πολιτισμού που είναι αρμόδια κατ' ουσίαν. Ο κύριος Ωραίο. Σας ευχαριστώ. Συμμερίζομαι κι εγώ πλήρω τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα της κυρίας Δελή. Και θα ήθελα να υποβάλω μία πρόταση. Ο εθελοντισμός πολύ συχνά εκδηλώνεται μέσω των σωματείων και των συνεταιρισμών, ιδιαίτερα στη Γαλλία, υπάρχει ε, τέτοιος ιστός ε, συνεταιριστικός πολύ πυκνός και πολύ συχνά τα σωματεία και οι σύλλογοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, ιδιαίτερα όταν είναι επιλέξιμα για κρατικές επενδύσεις και οι πρόεδροι αυτών των συλλόγων που πολλές φορές είναι θελοντές ε, εκτίθενται μερικές φορές και υφίστανται και διώξεις. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε ήδη από τώρα να προτείνουμε μια σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού, μια σύσταση ε, προς όλα τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν επιμελητήρια του εθελοντισμού, όπως υπάρχουν τα εμπορικά επιμελητήρια, τα γεωργικά, τα βιοτεχνικά, τα βιομηχανικά. Να υπάρχουν ειδικά επιμελητήρια εθελοντισμού που θα παρέχουν στους εθελοντές και δικαστική αρρωγή, αλλά και τεχνική υποστήριξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λογιστική διαχείριση. Γιατί εκεί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι έτσι θα βοηθούν πολλοί σύλλογοι και σωματεία που είναι οι κύριοι φορεί του εθελοντισμού σε πολλέ χώρε. Σα ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλον κανέναν κανένα θελοντή για το λόγο. Οπότε, μήπως θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στις συγκεκριμένες ερωτήσεις της κυρίας Κάθριν Μπέργκερ. Γιατί για τα υπόλοιπα θα συλλέξει όλες τις ε, απόψεις η συγκεκριμένη και θα επανέλθουμε τον Νοέμβριο στη συζήτηση. Α, παρέλειψε έναν ομιλητή, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την πρόταση αυτή. Είναι πραγματικά εξαιρετική ιδέα, γιατί πιστεύω ότι ο εθελετισμός όντω είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι και πολιτισμικό ζήτημα, το οποίο στην κεντρική Ευρώπη έχει πολύ μεγάλες ιστορικές ρίζες. Η εμπλοκή των νέων και όλα τα υπόλοιπα φυσικά συνεπάγονται ε, μεγάλη εξοικονόμηση σπόρων Και ξέρετε, σας λέω γιατί τα 14 μου συμμετέχω σε εθελοντική οργάνωση της Αυστρίας. Και γι' αυτό λοιπόν προχωρώ στο εξή αίτημα. Να μην ε, παραβλέπουμε τη διάσταση της ε, σωστής εργασιακής ε, κατάστασης, γιατί βλέπουμε στην Αυστρία ότι σε μεγάλες εθελοντικές παρεμβάσεις, επεμβάσεις στην Ελλάδα και στην Νότια Ευρώπη είναι έντανη και υπάρχει ένταση γιατί δεν χαίρονται όλοι οι εργοδότες αν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος τους αφιερώνει ένα, ε, μία μέρα για παράδειγμα στην πυροσβεστική για την καταπολέμηση των πλημμύρων. Υπάρχουν λοιπόν τα προβλήματα αυτά και να το ε, διευκρινίσουμε ότι δεν είναι όλοι φιλικά και θετικά διακείμενοι. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι εργατικές διατάξεις να ισχύουν καθολικά και γενικά. Thank you Σας ευχαριστώ. Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Αν θα μπορούσατε λοιπόν να απαντήσετε στη μία αυτή ερώτηση. Μία απάντηση μόνο στην ερώτηση της κυρίας Μπέργκερ. Καλώς, θα είμαι συνοπτική. Σας ευχαριστώ θερμά καταρχήν για τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας που εμπλουτίζουν τη συζήτηση και θα φροντίσω να αντικατοπτριστούν στην γνωμοδότησή μου. Όντως, ο προϋπολογισμός δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει σίγουρα να αναγνωρίσουμε το έργο των εθελοντών και σε ό,τι αφορά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, δεν είναι και πολύ σαφή τα πράγματα ακόμη. Πιστεύω ότι θα πρέπει ήδη να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της υιοθέτηση της απόφασης, γιατί το 2011 θα έρθει πολύ γρήγορα, οπότε καλύτερα να έχουμε γκρίνει τα κονδύλια. Καλώς, ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό αγαπητοί συνάδελφοι και προχωρούμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε προσκεκλημένο τον δόκτωρα Φαμπρίτσιο Μπάρκα, να σας ε, ενημερώσω καταρχήν ότι στα πλαίσια της ε, διαρκούς συζήτησης για την πολιτική συνοχής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκάλεσε τον κύριο Μπάρκα, τον δόκτωρα Μπάρκα, να εκπονήσει ανεξάρτητη έκθεση αξιολογώντας ε, την πολιτική συνοχής και υποβάλλοντας προτάσεις για τη μελλοντική μεταρρύθμιση της πολιτικής αυτής. Συνολικά οργανώθηκαν οκτώ ακροάσεις προκειμένου να εκπονηθεί αυτή η ανεξάρτητη έκθεση. Ήταν εκτενέστατες οι διαδικασίες. Σήμερα είναι μαζί μας ο Δόκτωρ Φαμπρίτσιο Μπάρκα για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του και να έχει μια ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής μας. Έχετε το λόγο κύριε Μπάρκα. Έχετε την πολυτέλεια του χρόνου. Όσο χρειάζεται για την παρουσίασή σας μπορείτε να τον έχετε. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που έχω την ευκαιρία να μιλήσω μπροστά στο δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα της Ευρώπης. Ένα σώμα το οποίο εξετάζει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχή, όπως συμπεραίνει η έκθεση, χρειάζεται μεταρρύθμιση. Θα μιλήσω αγγλικά γιατί η έκθεση είναι ούτως ή άλλως συνταγμένη στα αγγλικά και μου είναι πιο εύκολο. Yeah, okay, fine. Okay. actually, the, the only title, the only title of Ο μόνος τίτλος από την παρουσίασή μου που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν ο πρώτος. Η παρουσίασή μου ξεκινάει με το Back to the origin, πίσω στις ρίζες. Θα ξέρετε καλύτερα από μένα ότι η συνθήκη που χρόνει την Ένωση να επιδιώξει την ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εδαφικές επιπτώσεις και τον σχεδιασμό, τον καλύτερο σχεδιασμό της πολιτικής συνοχής. Ξέρετε ότι η πολιτική αυτή ενισχύθηκε τη δεκαετία του 70 και του 80 με στόχο να δώσει στους Ευρωπαίους πολίτες και σας θυμίζω εδώ την παρουσίαση του George Thompson του 73 ότι αναντήρητα η κοινή θέληση όλων να βοηθήσουν κάθε κράτος μέλος να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των πολιτών του ιδίω όπως συνεχίζει στην έκθεσή του, να διαθέσουμε που να αξιοποιούνται καλύτερα. Αυτό είναι ένα οικονομικό στόχο σε μια πρώτη φάση. Μιλάμε για αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα. Συνεχίζει όμω ο Τζορτ Τόμψον ότι θα πρέπει να γεφυρώσουμε τα χάσματα στι ε, συνθήκε διαβίωση. Αυτό είναι ένα κοινωνικό στόχο, ο οποίος υπονοεί την ισότητα, την κοινωνική συμμετοχή. Εδώ λοιπόν οι στόχοι ήταν πάντοτε ε, αυτή εξ αρχή οικονομική και κοινωνική. Γιατί όμως σα θυμίζω τέτοια πράγματα προφανή, διότι έχει γίνει η έννοια αυτή πλέον αμφιλεγόμενη. Η έκθεση υπονοεί ότι υπάρχουν παρανοήσεις για, την, ε, για τους στόχους της πολιτικής συνοχής και αυτή η παρανόηση παρεμποδίζει και την αποτελεσματικότητά της. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι ένα εργαλείο για την οικονομική διανομή πόρων μεταξύ των κρατών Δεν είναι μεταφορά κονδυλίων ε, ο στόχος της κοινωνικής της πολιτικής συνοχή. Η έκθεση λέει ότι αν αυτό ήταν ο στόχο, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε την πολιτική συνοχή, αλλά ένα ταμείο εξιστάθμιση. Με ομοσπονδιακό, ομοσπονδιακό ή τελείω ομοσπονδιακό χαρακτήρα. Με αυστηρού ελέγχου και μεταφορά κοντιλίων, χωρί διαδικασίε. Κανένα πρόβλημα. Σούπερα απλούστευση. Αλλά γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Διότι ο στόχο τη πολιτική συνοχή δεν είναι η επανακατανομή των κονδυλίων. Ο στόχο είναι η ανάπτυξη και μια αναπτυξιακή πολιτική που στοχεύει την ισότητα για τους δικαιούχους, την ίση κατανομή των πόρων και την κοινωνική συμπερίληψη μέσω της ε, ανακατανομής των κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών. Οπότε αμέσως τίθεται το ερώτημα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει αναπτυξιακή πολιτική. Με συγχωρείτε που ε, σας θυμίζω αυτά τα προφανή στοιχεία, αλλά εδώ υπάρχουν επικριτικά σχόλια και έλλειψη συνένεση πολλέ φορέ για αυτή την πολιτική, οι οποίε παρακολύουν την αποτελεσματικότητά της και την επιτυχία της. Η έκθεση εξετάζει το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, ιδίω στις ΗΠΑ. Ε, καμία ένωση κρατών με ενωπημένη αγορά και στο εργατικό δυναμικό και στα αγαθά, δεν μπορεί να μην έχει μια αναπτυξιακή πολιτική, η οποία να επιτρέπει στου πολίτε τη να υποφελούνται από τα πλεονεκτήματα τη αγορά και να αντιμετωπίζουν και του κινδύνου τη αγορά. Είναι τόσο απλό. Ήταν ε, και σαφές για τους ε, ιδρυτές της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Τώρα, οι προσδοκίε των πολιτών για πρόσβαση στην αγορά με ίσε ευκαιρίε είναι κάτι που οι προσδοκίε αυτέ δεν ικανοποιούνται πάντοτε. Οι πολίτε πολλέ φορέ θα έχουν αντιρρήσει για την κυκλοφορία των εργαζομένων, για την απελευθέρωση, για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην έχει εκμεταλλευτεί πλήρω όλε τι ευκαιρίε που τη έχουν δοθεί και γι' αυτό να υπάρχουν αντιρρήσει για την απελευθέρωση. Η έκθεση λοιπόν μελετά το τι συμβαίνει στι ΗΠΑ και το Ομοσπονδιακό Προπολογισμό υπολογισμό και βρίσκεται η αναπτυξιακή πολιτική των ΗΠΑ μοιάζει πολύ με τη δικιά μα. Απλώ είναι 3,5 φορέ μεγαλύτερη από ό,τι σε εμά. Είναι λογικό αυτό γιατί και η χώρα ίδια είναι πολύ μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά με τι ίδιε ιδέε. Στεγαστικέ παρεμβάσει, κοινωνικέ παρεμβάσει, εκπαίδευση, γέφυρε, υποδομέ, ε, στήριξη των επιχειρήσεων, περιβάλλον. Όμω, τι αναπτυξιακή πολιτική και εδώ είναι η τελευταία θεωρητική ερώτηση που θα θέσω πριν περάσω στην ουσία. Ποια είναι η κατάλληλη πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δύο μοντέλα που προωθούνται και θα προωθούνται και στο άμεσο μέλλον. Το ομοσπονδιακό είναι το πρώτο. Το ομοσπονδιακό και το μεακό όπου σε ομοσπονδιακό επίπεδο ένωση δημιουργείται ένα σύνολο κονδυλίων για την κοινοτομία, για τη μεταφορά άλλο, για τι κλιματικέ αλλαγέ, για την κοινωνική συμπερίληψη, για την απασχόληση, για τι ε, λαστασφάλειε και το καθεξή. Αυτά τα ταμεία λοιπόν ε, από το Ομοσπονδιακό Σώμα, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν υπάρχει προκαθορισμό των κονδυλίων. Αυτό είναι ο πρώτο τρόπο. Ο δεύτερο είναι ένα πολυτομεακό ταμείο το οποίο δεν ε, διαιρείται σε τομείς αλλά σε κράτη και περιφέρειες μέσω συμβάσεων συμβάσεων ε, μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών. Βάσει αυτών των συμβάσεων οι δωρεές προς τα παροχές προς τα προγράμματα και τα σχέδια των κρατών μελών γίνονται βάσει του σεβασμού συγκεκριμένων αρχών. Αυτό είναι το δεύτερο μοντέλο. Οι ΗΠΑ ακολουθούν το πρώτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί το δεύτερο. Και υπάρχουν δύο λόγοι για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση τονίζει ότι οι λόγοι αυτοί ισχύουν περισσότερο από ποτέ σήμερα. Γιατί πρώτον αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Η αναπτυξιακή θεωρία δεν είναι κάτι που θα αναπτύξω εδώ, δεν υπάρχει χρόνο γι' αυτό, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια τα λέει και η έκθεση. Έχουμε περάσει προ το δεύτερο μοντέλο στην αναπτυξιακή θεωρία. Έχουμε μάθει από τα λάθη της Παγκόσμιας Τράπεζας, από τα λάθη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από τα λάθη του ΟΣΑ. Υπάρχει λοιπόν ένα νέο παράδειγμα περιφερειακής πολιτικής, αναπτυξιακής πολιτικής, το οποίο υπονοεί με σαφήνεια ότι ο μόνο τρόπο να προχωρήσει κανεί είναι με μια πολιτική που λαμβάνει υπόψη τη γνώση και τι προτιμήσει των πολιτών που ζουν σε συγκεκριμένα μέρη, τόπου. Ο τρόπο να γίνει αυτό δεν είναι με μια πολιτική που ξεκινά από τι αρχέ και με τομιακή παρέμβαση πηγαίνει προ τα κατώτερα επίπεδα. Όχι. Οι Αμερικανοί φίλοι μα, όπω λέει κάποιο που γνωρίζω από την πόλη του Κάνσα, λένε ότι πολλέ φορέ στι αναπτυξιακέ πολιτικέ ε, το one size fits all, δηλαδή ένα μέγεθο κάνει για όλα αλλά το θέμα είναι και οι οικονομικοί λόγοι. Γιατί δεν επιλέγουμε την τομεακή ε, κατεύθυνση. Ο τομεα... Η τομεακή προσέγγιση είναι ανέφικτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικό μας μοντέλο είναι το μόνο το οποίο είναι συμβατό με την περιορισμένη δημοκρατική θεμητότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν θεσμικά όργανα στο υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο τα οποία να έχουν οργανισμού και να πηγαίνουν στο έδαφο μετά των κατομελών στην επικράτειά του, να στείλουν ε, τέντε και να αποφασίζουν πώ ακριβώ θα υλοποιείται η πολιτική. Αυτό μπορεί να γίνει σε 150 χρόνια από σήμερα. Σήμερα όμω δεν μπορεί να γίνει αυτό στι περιφέρειε, ε, ούτε θα ήταν συνεπέ με τι εθνικέ προσδοκίε των 100 μελών. Ο μόνο τρόπο λοιπόν να προχωρήσουμε για να επιτύχουμε του στόχου τη αναπτυξιακή πολιτική είναι με μια πολιτική όπου τα κράτη, οι περιφέρειε δηλαδή και οι επαρχίε έχουν τη δυνατότητα υλοποίηση ενώ τα κράτη-μέλη δίνουν απλώ τι κατευθυντηρίε γραμμέ. Πέραν τώρα αυτού, ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι όλα αυτά είναι αρκετά σύγχρονα. Κάποιοι λένε ότι είμαστε παροχημένοι στην προσέγγιση μα. Όχι. Αυτό είναι ο σύγχρονο τρόπο καθορισμού του ε, προπολογισμού. Και εδώ έχω μια σειρά από λόγου. Δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτού. Έχω και άλλα να σα αναπτύξω. Απλώ να τα αναφέρω πολύ σύντομα. Γιατί σήμερα θα πρέπει να ανανεώσουμε τι προσπάθειέ μα για να κάνουμε πιο αποτελεσματική την πολιτική συνοχή. Πρώτα απ' όλα γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτε σήμερα δεν λαμβάνουν του καρπού τη πολιτική αυτή. Δεν αισθάνονται ότι έλεγε, όπως έλεγε και ο Τζορτ Τόμψον, ότι δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης της κοινή βούλησης. Αμφισβητείται η κοινή βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παντού. Και αυτό φαίνεται όποτε ψηφίζουν και αναλαμβάνουν δράση οι πολίτες. Ή, όταν δεν ψηφίζουν και απέχουν από τις εκλογές. Η πολιτική λοιπόν συνοχής σήμερα δεν γίνεται αντιληπτή ως ισχυρή ώστε να ωφελήσει τους πολίτες έπειτα. Υπάρχουν και διάφορες παρανοήσεις όπως είπα προηγουμένως, οικονομική ανακατανομή κονδυλίων Έπειτα είναι η σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία μας υποχρεώνει με περισσότερο, με ανανομένες και εντατικότερε προσπάθειες να δράσουμε, διότι τα δημόσια κονδύλια πλέον δεν είναι πολλά και θα πρέπει να, να παράγουμε αποτελέσματα, να δώσουμε καρπούς, γιατί έχουμε λιγότερα. Και κατά δεύτερον, επειδή η κρίση προκαλεί και απαιτεί προσαρμογέ των περιφερειών βιομηχανικού πλέον επίπεδου. Οι επιχειρήσει και οι βιομηχανίε παντού γνωρίζουν τριγμού. Χρειάζονται λοιπόν προσαρμογέ και χρειάζεται εδώ η πολιτική και τα εργαλεία τη αγορά. Και υπάρχει και ένα πολιτικό επιχείρημα εδώ, ένα πολιτικό λόγο και μετά θα προχωρήσω, θα σα πω τι αλλαγέ πρέπει να γίνουν. Σε σύγκριση με το τι συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια, το θέμα της πρόθεσης της Ευρώπης των λαών, αυτό έχει ξανάρθει στο προσκήνιο. Εάν δούμε τη σειρά προτεραιοτήτων του Προέδρου Μπαρόζο που πήρε την ψήφο της πλειοψηφίας από εσά, μας καλεί να έχουμε ίση μεταχείριση για τους Ευρωπαίους πολίτες και αυτό να γίνει πραγματικότητα. Ή επίση καλή να γίνει χρήση των, να, ασκήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτε τα δικαιώματά του ω Ευρωπαίοι πολίτε κατά τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούν τα εθνικά του δικαιώματα ω εθνικοί πολίτε. Ο μόνο τρόπο να, να καλυφθούν αυτέ οι προσδοκίε, να ικανοποιηθούν, είναι η αναπτυξιακή πολιτική. Και η μόνη εφικτή αναπτυξιακή πολιτική για την Ευρώπη είναι αυτή που θα βασίζεται στου τόπου, δηλαδή η πολιτική συνοχή. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε, να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχή. Η έκθεση, αφού αναλύει μέσα από μία μακροσκελή συζήτηση και με τη συμμετοχή 40 ακοδημαϊκών καθηγητών πανεπιστημίων, ε, ε, συμμετεχόντων από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών, ε, από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, έλεγαν ότι η μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής συνοχής πρέπει να έχει δύο σκέλη. Το πρώτο το έχω συζητήσει. Έπειτα πρέπει να υπάρχει και μια πολιτική διάσταση. Θα πρέπει να γίνει πιο σαφέ ότι η κοινωνική συνοχή είναι μια πολιτική για την ανάπτυξη και πρέπει να έχει δύο στόχου. Πολύ διακριτού μεταξύ του, αλλά δύο, δύο και όχι έναν. Την αποτελεσματικότητα και την ισότητα, την κοινωνική συμπεριλήψη και την μείωση τη ε, μη χρήση των πόρων. Υπάρχει μια σημαντικότατη κοινωνική διάσταση εδώ. Δεν θα αναλύσω όλε τι λεπτομέρειε γιατί θα μιλήσω για πάρα πολλή ώρα, αλλά θα επανέλθω στην συγκεκριμένη κοινωνική διάσταση. Όμω, γιατί η κοινωνική διάσταση τη πολιτική συνοχή είναι ιδιαίτερα σοβαρή Α περάσουμε στο δεύτερο σκέλο αυτή τη συνολική μεταρρύθμιση. Σα ε, τα είπα γιατί η έκθεση είναι και τόσο περίπλοκη και έχει τόσε λεπτομέρειε. Σα τα λέω κάπω συνοπτικά. Αλλά θέλουμε εδώ να δώσουμε πρακτικέ συμβουλέ και ανακεφαλαιώνεται αυτό και στο διάγραμμα. Στο διάγραμμα όπου, όπω και η έκθεση στο τέλο τη, λέει ότι ο πυρήνα, η ουσία τη έκθεση είναι ένα κύκλο. Αλλά Υπάρχουν δύο ακόμη συστατικά που λείπουν και τα οποία είναι απαραίτητα. Τα οποία βρίσκονται στο κάτω μέρο του διαγράμματο. Για να γίνουν όλα αυτά να πετύχουν οι διαπραγματεύσεις είναι η συγκέντρωση σε βασικές προτεραιότητες και οι συμβάσεις με στόχο, με προοπτική τα, τα αποτελέσματα και επίσης η επικέντρωσή μας στη γνώση. Για να εργαστούμε λοιπόν σωστά πρέπει να ενισχύσουμε την Επιτροπή να ενισχύσουμε επίσης τον πολιτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Αυτό είναι ο ρόλος μας. Για να πετύχουν όλα αυτά πρέπει το σύστημα διαπραγματεύσεών μας δραστικά να το αναθεωρήσουμε. Και θα το σχολιάζω και αυτό εντάχει για να περάσουμε μετά τις ερωτήσεις. Συγκέντρωση. Η έκθεση λέει ότι τα δύο τρίτα όλων των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε τρεις ή τέσσερις βασικές προτεραιότητες το πολύ αλλά θα πρέπει να υπάρξει σαφή ουσιαστική συγκέντρωση, όχι συγκέντρωση όπω αυτή που εννοούσαμε με τη στατική τη Λισαβόνα, όπου στο τέλο όλε οι δυνατέ χρήσει τελικά επιτρέπονταν. Αντικείμενο συμβάσεων, διαπραγματεύσεων, γιατί η ατζέντα τη Λισαβόνα ήταν τόσο ευρεία που κάλυπτε τα πάντα. Εδώ θέλουμε λίγε βασικέ προτεραιότητε. Ποιε, λόγου χάρη. Η έκθεση λέει ότι δεν μπορούν οι τεχνοκράτε να καθορίσουν εδώ ή να κάνουν προτάσει, πρέπει να υπάρξει πολιτικό διάλογο. Η έκθεση απλώ δίνει ιδέε για τη συζήτηση. Οι προτάσει λοιπόν που γίνονται είναι για το στόχο τη αποτελεσματικότητα. Καινοτομία, προφανέ. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την καινοτομία. Γιατί θα πρέπει η καινοτομία να είναι μια βασική προτεραιότητα. Και η προσαρμογή στι κλιματικέ αλλαγέ. Όχι αναχέτηση, όχι μετριασμό των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Γιατί εκεί περιμένουμε τις επιπτώσεις. Εδώ θέλουμε να είμαστε αποδοτικοί και στο κοινωνικό σκέλος βασική πρόταση είναι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης, δηλαδή όχι μόνο υπηρεσίε για τους μετανάστες, αλλά υπηρεσίε για τους ανθρώπους όπου κατοικούν οι μετανάστες, υπηρεσίε για τους ανθρώπους, για τις περιοχές μάλλον από όπου προέρχονται οι μετανάστες. Θα πρέπει εδώ να ασχοληθούμε με το θέμα τη ποιότητα με, με τις βασικές προδιαγραφές διαβίωσης όλων των πολιτών. Γιατί όλου μα αφορά η μετανάστευση. Ή τα παιδιά που, όπως ξέρετε, είναι ήδη στο κέντρο της συζήτησης για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και εκεί μας αφορά το θέμα της μετανάστευσης. Και υπάρχουν και άλλες δύο επιλογές, αλλά όλα αυτά τα συζητήσετε εσείς. Δεν είναι δική μου δουλειά να τα αποφασίσω, δική σας, δικό σας έργο είναι. Οι δεξιότητες, η προσαρμογή των δεξιοτήτων και των προσόντων. Η έκθεση λοιπόν τι λέει, μην πάρετε έναν τομέα, τις μεταφορές λόγου χάρη, ή την εκπαίδευση ή τα κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, αλλά ζητήματα που αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες, αυτά που τους απασχολούν και έπειτα να επικεντρώσουμε τις πολιτικές μας στο τι ε, χρειάζεται να γίνει βάσει αυτών των θεμάτων. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση. Η δεύτερη είναι το τι γίνεται με τις συμβάσεις. Η ουσία της πολιτική αυτής είναι να επιτρέψει τη λειτουργία της επικουρικότητας. Εάν δεν υπάρχει αρκετή επικουρικότητα, η πολιτική αυτή χάνει το νόημά τη. Δεν επιτρέπουμε στου πολίτε να γνωστοποιήσουν τι προτιμήσει του. Εάν υπάρχει όμω υπερβολική επικουρικότητα, καταλήγουμε να ζούμε σε περιοχέ απομονωμένε, χωρί κανόνε. Χάνουμε την ευρωπαϊκή διάσταση και τι ευρωπαϊκέ αρχέ και αξίε. Χρειάζεται λοιπόν ισορροπία μεταξύ τη ευρωπαϊκή αρχή από τη μια και τη πραγματική κινητοποίηση των τοπικών πόρων από την άλλη. Αυτό γίνεται βάση των συμβάσεων. Αυτό θα είναι το στρατηγικό μας πλαίσιο. Για τα λειτουργικά προγράμματα. Η έκθεση λέει ότι σήμερα οι συμβάσει επιβαρύνουν τα κρατημέλη και τις περιφερειές με τεράστιες διαδικαστικές απαιτήσει. Θα πρέπει λοιπόν να είναι περισσότερο ελεύθερες οι χώρες να αποφασίζουν μόνες πώς να φέρουν εις πέρα σε αυτέ τι διαδικασίε και να δεσμεύονται στις συμβάσει τους για δύο πράγματα επί τη ουσία. Αν επιλέξουν τη μετανάστευση. Να πούν ποια είναι τα αποτελέσματα που επιδιώκουν, λόγου χάρη. Δηλαδή, οι μαθηματικές δεξιότητες των παιδιών στις αστικές περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ε, προσέλευση μεταναστών να μην ε, μειωθούν λόγου χάρη. Θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά με αριθμητικά στοιχεία, να σημειωθούν στόχοι συγκεκριμένοι. Αυτό έχει γίνει ως προσπάθεια στην πολιτική συνοχή, αλλά δεν έχει πετύχει. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, δεν έχουμε καλούς δείκτες για αυτή την πολιτική. Δεν τα έχουμε συζητήσει ποτέ επαρκώς. Και όπως σας έχω πει, δεν μου ζητήθηκε ποτέ από το Ευρωκοινοβούλιο ε, από τότε που ανέλαβα στο νότο τη χώρα μου ευθύνε για αυτή την πολιτική. Εγώ ήμουν πάντοτε στη διάθεσή σα, αλλά και δεν έφταγε και το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι το σύστημα τέτοιο που δεν επιτρέπει την επικοινωνία μα. Δεν ζητούνται ποτέ οι πολιτικοί θύνοντε. Δεν του ζητάτε να έρθουν να συζητήσουν. Πάντω έστειλε ένα σύντομο μας στη Βουλή των Λόρδων γιατί δέχτηκα πολλά επικριτικά σχόλια. Σε αυτό το πλαίσιο, πρώτα απ' όλα πρέπει να θέσουμε στόχους με συγκεκριμένα αποτελέσματα και δεύτερη απέτηση που πρέπει να έχουν χώρε είναι το θεσμικό πλαίσιο. Μια κουβέντα γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα λέει η Επιτροπή στι περιφέρειες και τι επαρχίε τι θεσμικά όργανα να δημιουργήσουν. Αλλιώ παραβαίνουμε την επικορικότητα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο κανόνων ή αρχών. Εκπαίδευση λόγου χάρη. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα χωρί καλή αξιολόγηση, χωρί αξιολόγηση των προσόντων, για την ε, πρόσληψη δασκάλων. Ένα λογικό σύστημα αμοιβή των δασκάλων. Δεν υπάρχει λόγο να δαπανούμε κονδύλια και δαπανούνται πάρα πολλά για το εκπαιδευτικό σύστημα, ούτω ή άλλω. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να έχει την εξουσία και να έχει και την ευκαιρία, οι αρχέ, τι οποίε όλοι έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μα, γιατί οι περιφέρειες ε, και μέσω του όσα έχουν ε, συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτέ τι προσπάθειε. Εάν δεν συμφωνήσουμε λοιπόν και αν δεν επιτρέψουμε στην Επιτροπή όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγο να προχωρήσουμε. Θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι, το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο, να ξέρουν προ ποια κατεύθυνση κινείται μια χώρα και αν είναι σωστή ή όχι. Θα πρέπει να υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία. Οι στόχοι να είναι ποσοτικοί. Εάν μια χώρα που δεν επιτυγχάνει τα επιτελέσματά τη, εντάξει, μπορεί να μην πρέπει να τη επιβάλλουμε κυρώσει, αλλά την πιέσουμε να πάει προ τη σωστή κατεύθυνση, να μα δώσει εξηγήσει Εάν οι εξηγήσει είναι ικανοποιητικέ, θα μπορούσε να εκδώσει μια σύσταση η Επιτροπή. Αν δεν ακολουθηθεί η σύσταση, βλέπουμε. Αλλά το τελευταίο μέρο του κύκλου, και εδώ προχωρώ προ το τέλο, είναι η κινητοποίηση των παραγόντων και η μάθηση. Θέλουμε συγκέντρωση των πόρων, ωραίο είναι αυτό, ωραίο είναι να έχουμε καλύτερε συμβάσει, αλλά αν δεν βελτιώσουμε την κινητοποίηση των ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο, χάνουμε το στόχο τη πολιτική αυτή. Τι σημαίνει αυτό, δύο πράγματα. Ότι πρέπει να δώσουμε πίσω ένα πολύ μικρό ποσό κονδυλίων, πόρων στην Επιτροπή, για να κάνει καλύτερα κάποια από αυτά που ήδη κάνει τα τελευταία χρόνια. Πειραματισμό δηλαδή και καινοτομία. Πρέπει να έχει και κάποια... κάποιου πόρου για να το κάνει αυτό η Επιτροπή. Δεν χρειάζεται πολλά, αλλά λίγα για να μπορεί. Και έπειτα η αξιολόγηση τύπου Είχα πει ότι δεν θα μιλήσω για πάρα πολλή ώρα και τελικά θα αναγκαστώ να γίνω σύντομο. Χρειαζόμαστε χρόνο, ε, χρονομετρικές αναλύσεις, χρειαζόμαστε μαθηματικές μεθόδους. Απλές υπάρχουν, δεν είμαι ο ίδιος στατιστικολόγος, αλλά έχω ασχοληθεί με στατιστικά δεδομένα και γνωρίζω το μαύρο κουτί κάποιων μεθοδολογιών. Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε έγγραφα με αξιολογήσει που στο τέλο μα εξηγούν ότι χρησιμοποίησαν μεθοδολογία την οποία δεν καταλαβαίνει κανεί και μα λένε τελικά μια πολιτική πέτυχε ή όχι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν τώρα μεθοδολογίε, ιδίω ένα σύστημα που ονομάζεται μελέτη αντικτύπου, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προγράμματα και σχέδια με πολύ απλό τρόπο. Πολύ απλά μπορεί να πει κανεί ότι εδώ έχουμε μια ομάδα εταιριών, επιχειρήσεων ή πολιτών ή δικαιούχων που έλαβαν εκπαίδευση ή δικαιούχων που δεν έλαβαν εκπαίδευση. Α δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα. Απλούστατη μέθοδο. Έτσι, η, κοινωνική, η πολιτική μάλλον συνοχή υιοθετεί μια τέτοια μέθοδο και μπορεί να αξιολογηθεί. Εάν λέμε λοιπόν ότι θέλουμε ένα στόχο συν 25% για την εκπαίδευση, α το εφαρμόσουμε αυτό. Το έμαθα αυτό συνεργαζόμενο με την Επιτροπή εδώ και χρόνια. Και είχα συζητήσει με τι υπηρεσίε αξιολόγηση και επειδή είχα εγώ ίδιο τη δυνατότητα και επειδή μου ζητήθηκε. Και όχι μόνο μπορούμε έτσι μια επταετία αργότερα να γνωρίζουμε αν κάτι τελικά υλοποιήθηκε ή όχι, αλλά έχει και ένα αποτέλεσμα προ την πειθαρχία αυτό, διότι οι προγραμματιστέ αυτοί που υλοποιούν το πρόγραμμα, καταλαβαίνουν και συμμορφώνονται με το ότι πρέπει να πετύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Κάνουν καλύτερα τη δουλειά του. Ο στόχο δεν είναι απλώ να δαπανούν κονδύλια, να οργανώνουν συναντήσει πρέπει να στοχεύουν και σε ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα για τους δικαιούχους. Και εδώ δεύω προς το τέλος, γιατί μέχρι τώρα σας έλεγα πράγματα προφανή. Εδώ έχετε τεχνοκρατικές προτάσεις και έτσι θα μείνουν, εκτός και αν κάνουμε δύο διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα ενίσχυση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Γενικών Διευθυντών που είναι υπεύθυνη, διότι εάν συγκεντρώσουμε τα κονδύλια σε βασικέ προτεραιότητε όπω η μετανάστευση, τα κάτι μέλη και οι περιφέρειε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στι Βρυξέλλε δεν υπάρχουν μόνο δύο εξαίρετοι συνεργάτε που εργάζονται για το θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν 21. Ότι ο καθένα έχει τι καλύτερε δεξιότητε, μπορεί να εργαστεί με τον καλύτερο τρόπο για να δώσει τεχνική στήριξη, κατανόηση και θα συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή ακόμη και όταν έχει απέναντί μα κάποιον σκληρό διαπραγματευτή η Επιτροπή. Εδώ υπάρχουν εθνικά ενδιαφέροντα, τα οποία και εμά πολλέ φορέ μα έφυγαν, ε, αλλά αναγκαζόμαστε να παραδεχτούμε ότι έχει δίκιο ο διαπραγματευτή τη Επιτροπή. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολύ σκληρού διαπραγματευτέ, οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν και χρειαζόνται πολύ ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση και Περιφερειών και των υπόλοιπων τομεακών γενικών διευθύνσεων. Και τέλο είναι η πολιτική έλεγχη και ισορροπίε. Η πολιτική αυτή μεταρρύθμιση που προτείνεται υπονοεί ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη διακριτική ευχαίρεια τη Επιτροπή, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σωστό αυτό. Θα μπορεί να πάει μια Επιτροπή σε μια χώρα και να τη πει χώρα, έχετε το σωστό θεσμικό όργανο ή όχι. Ή θα σα αναστείλω για ένα χρόνο. Και θα δούμε αν θα δημιουργήσετε το κατάλληλο θεσμικό όργανο ή όχι. Αυτό αυξάνει τη διακριτική, αυξάνει τη διακριτική ευχαίρεια τη Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε όμω ελέγχου και αξιολογήσει από το, και από αυτό από την πλευρά των άλλων δύο θεσμικών οργάνων. Και όχι μόνο το απαιτεί αυτή η διαδικασία, αλλά σε ένα τέτοιο σκηνικό θα είχαμε σαφέστερους στόχους ε, και τη δυνατότητα για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να έχουν και κάτι να συζητήσουν. Να πούν πηγαίνει σωστή κατεύθυνση μια χώρα ή όχι. Σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει. Όχι τους στόχους που κάποιος άλλος έξωθεν τις έχει επιβάλει. Να λοιπόν η συμμετοχή του Συμβουλίου στην ε, πολιτική συνοχή. Εδώ εκμεταλλευόμαστε και το άρθρο 275 της συνθήκης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωκοινοβούλιο να ετοιμάζει έκθεση αξιολόγηση σχετικά και να αποφαίνεται για τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής, ε, τα οποία θα γίνουν αναπόφευκτα στο μέρος των Εύρου του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 275. Το αντικείμενο συζήτηση λοιπόν του Ευρωκοινοβουλίου, του δικού σα σώματο. όχι μόνο τα σταλίε και χρονικές καθυστερήσει και έγκαιρη δαπάνη, και τέλος, χρειάζεται ένα χρονοδιάγραμμα, όπως για κάθε πρόταση, προφανώς Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσω. Το 2010 κιόλα. Δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνο για τη μεταρρύθμιση, αν θέλουμε να πετύχει. Εδώ θα χρειαστούμε τουλάχιστον ένα-δύο χρόνια εντατικών συζητήσεων για να καταλήξουμε στι βασικέ προτεραιότητε, οι οποίε πρέπει να προκύψουν από διαβουλεύσει, από πολιτικό διάλογο στα κράτη-μέλη και τέλο θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία. Τι προτείνετε εδώ, ότι όχι όπω κάνουμε σήμερα, το γνωρίζετε εσεί πολύ καλά. Πρώτα συμφωνούμε για το χρήμα, και εννιά μήνες μετά για τους στόχους και τους κανόνες. Ένας αριανός, αν έρχονταν από τον Άρη, δεν θα καταλάβαινε γιατί μια ομάδα ανθρώπων πρώτα προβλέπει πώς θα κατανέμει τα κονδύλια και μετά προβλέπει τη σύμβαση για το πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλια και για ποιους στόχους. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη λοιπόν παράλληλη εξέταση των θεμάτων αυτών. Αλλιώς οι εγωισμοί των κρατών προκύπτουν όταν ε, αποφασίζεται η κατανομή των κονδυλίων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε αρχικά ελεύθεροι στις επιλογές μας και να μην περιμένουμε 6-9 μήνες όπου βλέπουμε τη διάβρωση των στόχων, τη διάβρωση των κανόνων και των κανονισμών να συμβαίνει. Εδώ βέβαια χρειάζονται και πολιτικοί συμβασμοί και παραχωρήσεις και είναι σαφής ο, σαφ... ο σημαντικότατος ρόλος που εσείς στο Ευρωκοινοβούλιο έχετε να διαδραματίσετε εδώ. Ευχαριστώ. Η πρόεδρο. Προβλεπόταν συζήτηση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα σχόλιά σα με τι ερωτήσει σα και μετά θα ομαδοποιούμε τι ερωτήσει και θα απαντάτε. Σέτελ. Um, ευχαριστώ. κυρία Σρόιντερ, Είμαι εντυπωσιασμένη που επιτέλους βγαίνετε και μιλάτε και αναφέρετε αυτές τις αλήθειες. Είπατε λοιπόν με σαφήνεια τα τελευταία πέντε έτη συνέβησαν σφάλματα και είναι σαφές ότι αυτή η πολιτική του earmarking την οποία επί χρόνια ε, καταδίκαζα την καταδικάσατε κι εσείς. Αυτό σήμαινε ότι χάθηκαν χρόνια. Αυτή η πολιτική, αυτή η ενσωματεμένη πολιτική συνοχής και θα μας βασανίσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε ότι οι περιφέρειες εκείνες οι οποίες χρειάζονται πιο πολύ τη βοήθεια δεν προχώρησαν καθόλου τότε προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επανάσταση, γιατί αυτό επιβλήθηκε στο Κοινοβούλιο, αυτή η εισαγωγή της πολιτικής του earmarking. Δεν το καταφέραμε. Δεν το καταφέραμε γιατί δεν το επιθυμούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελε οπωσδήποτε αυτό το earmarking. Αυτό που είπατε λοιπόν τώρα είναι να επιστρέψουμε στις ρίζες της πολιτικής συνοχής, στις αρχές της, βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας και εταιρικής σχέσης. σε όλα αυτά στα οποία απέδειξε αδυναμία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εξαιρετικό το μήνυμά σας. Είπατε να επιστρέψουμε και σε μια πολιτική η οποία καταδικάστηκε επί σειρά ετών. Το πείραμα λοιπόν αυτό ας μας διδάξει. Είχαμε τις ε, κοινοτικές πρωτοβουλίες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν ε, μικροσκοπικές αλλά τις αγαπούσαν όλοι, γιατί επέτρεπαν αυτά τα πειράματα, επέτρεπαν επιτόπου οι φορείς να συμμετέχουν στον προγραμματισμό. Έκαναν λοιπόν ε, τα πειράματα και ανέλαβαν και τη σχετική ευθύνη. Καταργήθηκε αυτή η πολιτική. Δεν ανανεώθηκε. Στην έκθεση σας φαίνεται σαφώς ότι πρόκειται για λάθος. Ξέρουμε ποια είναι οι δυναμίες. Γραφειοκρατία, υπερβολική επιβάρυνση μικρών φορέων. Αυτά τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν, ούτε εσείς τα επιλύσατε. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι οι μέθοδοι που υπήρχαν στις κοινοτικέ πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στις τελευταίες τρεις, Equal Leader και Interreg, θα πρέπει εκ νέου να εφαρμοστούν. Και καθίσταται σαφές ότι αυτή η αποκεντρωμένη διάσταση την οποία δεν αποδέχονται τα κράτη-μέλη παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τα σχετικά μέσα, δεν αξιοποιούνται και δεν ξεκίνησε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα κράτη-μέλη εκείνα όπου χρειαζόταν. Τα αφήσαμε ελεύθερα και είπαμε ότι α, δεν αναμειγνιόμαστε, δεν μπορούμε να αναμειχθούμε στα εσωτερικά των κρατών μελών και σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την έκθεσή σας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενθαρρυντική για μας, ε, ανθρώπους εγκεμένα που επί 20 χρόνια ασχολούμαστε με την περιφερειακή πολιτική. Να επιστρέψουμε στις ρίζες ε, της εταιρική σχέσης, της συνεργασίας και κυρίως επιστροφή προκειμένου ο κόσμος επιτόπου να είναι αυτός που δημιουργεί τα προγράμματα, να μην πρόκειται για δημιουργήματα των εθνικών κυβερνήσεων. Θα πρέπει να συνεχίζουμε λοιπόν τις συζητήσεις αυτές προκειμένου να καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα και να μην δημιουργήσουμε εκ νέου μια γραφειοκρατική διαδικασία όπως ήταν αυτή η διαδικασία του earmarking που ουσιαστικά απέτρεψε κάθε καινοτομία και είχε μηδενικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Κωνσταντσε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι την ίδια παρουσίαση, ακούσαμε. Είναι πραγματικά εξαιρετική η έκθεση, να το πω αυτό, και πραγματικά ενισχύονται πολλές μου ιδέες. Αλλά δεν τα άκουσα τα πράγματα όπως μας τα παρουσίασε η Ελίζαμπεθ τώρα πριν από λίγο. Και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Αν σωστά κατάλαβα κύριε Μπάρκα, αυτό που λέτε είναι ότι η συγκέντρωση θα πρέπει να υπάρξει συγκέντρωση σε συγκεκριμένε προτεραιότητε. Ποιε θα είναι αυτέ οι προτεραιότητε θα το κοιτάξουμε. Αλλά αυτό τι σημαίνει ότι απομακρύνεστε από το γεγονό ότι στο μέλλον, για παράδειγμα, μεγάλος, ε, μεγάλο με, με, ποσοστό των κονδυλίων θα δίνεται για τις υποδομές, για παράδειγμα. Σωστά. Καταλαβαίνω θα ήθελα όντως να γίνει αυτή η επικέντρωση στις προτεραιότητες, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό εννοείται με ένα μεγάλο αγώνα με τα κρατημέλη, για παράδειγμα. Ύστερα, κάτι που δεν κατάλαβα. Στην μελλοντική συνθήκη, στην συνθήκη της Λισαβόνας, ο τρίτος πυλώνας της πολιτικής συνοχής πέρα από την οικονομική συνεργασία και την ε, κοινωνική συνοχή αναφέρεται και η εδαφική συνοχή στη συνθήκη. Πώς φαντάζεστε εσείς ότι η νέα πολιτική συνοχή θα αλλάξει, ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει και θα έπρεπε να ακολουθήσει. Σύμφωνα με τα εφιστάμενα κριτήρια, αν τα ανάγουμε, ο πρώτος στόχος κάτω του 75% και ο δεύτερος στόχος κτλ. Με τα εφιστάμενα λοιπόν κριτήρια στην Ευρώπη των 15 δεν θα υπήρχαν σχεδόν καμία περιοχή στόχου 1 πλέον. Αυτό το καταδεικνύουν όλα τα στατιστικά στοιχεία. Ξέρω ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν την εντύπωση ότι στο μέλλον θα επικεντρώνουν όλα τα κονδύλια στις περιοχές στόχου 1, το οποίο θα σήμαινε ότι η κεντρική και βόρεια Ευρώπη δεν θα είχαν πλέον μέσα συνοχής. Πώς τοποθετήσετε εσείς, συμφωνείτε με αυτή την αντίληψη ή θα ήταν διαφορετική η προσέγγιση σας. Τρίτη ερώτηση. Για μένα η κοινωνική συνοχή η πολιτική συνοχή, συγγνώμη, δεν έχει να κάνει μόνο με τα τρία μέσα, με το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Περιφερειακό Ταμείο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και ανάπτυξη της υπαίθρου. Εσείς θεωρείτε ότι το τμήμα αυτό της ε, προώθησης της ευρωπαϊκής πολιτικής θα πρέπει να επανέλθει στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής ή τάσσεστε υπέρ της τρέχουσας διάκρισης που επικρατεί σήμερα. Ευχαριστώ, Κωνσταντσε, ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή. Τη έριξα και μια μάτια πριν ε, τη συνεδρίαση και ήταν λίγο διαφορετική η αντίληψή μου σε σχέση με την αντίληψη της συναδέλφου Σρόντερ. Εγώ θεωρώ ότι το earmarking ήταν μια πολύ καλή διαδικασία, γιατί αποτελεί εγγύηση για το ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα χρήματα του φορολογούμενου, δεν μπλέκουν σε διάφορες προβληματικές περιοχές. Έχουμε σαφείς στόχους και γυσμοί και οι καλές περιφέρειες, οι καλές ιδέες μπορούν να ζητήσουν τα κονδύλια αυτά. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια εγγύηση σωστών επενδύσεων. Αυτό ως μια πρώτη παρατήρηση. Με ενοχλεί κάπως η αντίληψή σας για την πολιτική διάρθρωσης. Είπατε ότι τα ανοιχτά σύνορα δεν είναι μόνο καλά. Αλλά πώς προκύπτει η ευημερία, να ρωτιέμαι. Η ευημερία προκύπτει όταν τα κράτη-μέλη ε, εμπορεύονται σε ανάλογο επίπεδο. Όταν ε, αγοράζει ένας Γερμανός ε, ένα Fiat από την Ιταλία γιατί πιστεύει ότι είναι καλό και το ίδιο κάνει και ο Ιταλός με μία BMW. Η πολιτική διάρθρωσής μας ήταν επί χρόνια επικεντρωμένη στην διευκόλυνση του εμπορίου αυτού σε χώρες που δεν είχαν αντίστοιχο επίπεδο. Στην εκπαίδευση, στην καινοτομία, στην έρευνα. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι αποτυχημένη αυτή η πολιτική. Νομίζω ότι απέδειξε την αξία της, γιατί βλέπουμε ότι όντως τα ποσοστά ανάπτυξης τα οποία προκλήθηκαν από την πολιτική συνοχή στις χώρες αυτές είναι σημαντικά και βλέπουμε επίσης και σημαντικές θετικές επιδράσεις και στις χώρες της δωρήτριες, αν θέλετε, που έδωσαν τα κονδύλια. Αυτό το καταδεικνύουν όλες οι μελέτες. Και επίσης με ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό που προτείνεται ως ε, μελλοντικές προτεραιότητες. Ε, ωραία, εντάξει, τα παιδιά, η εκπαίδευση, η μετανάστευση. Αλλά ξεχνάτε τα κλασικά μέσα. Την προώθηση της ε, ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας των θέσεων εργασίας. Είτε δεν κατάλαβα σωστά, είτε κινείστε προς μία κατεύθυνση την οποία εγώ προσωπικά θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνη. Δεν αποτελεί αυτό το μέλλον, θεωρώ, της πολιτικής συνοχής. Μία τελευταία παρατήρηση, μάλλον προτελευταία. Μου αρέσει το γεγονός ότι ως κριτήριο σας αρέσει το ΑΕΠ, η μέτρηση δηλαδή, ε, μάλλον το καθάριστο κοινωνικό προϊόν ως ε, μέτρο σύγκρισης. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Τι εννοείται Συμβούλιο για την Πολιτική Συνοχής. Θεωρείτε ότι τα κράτη-μέλη πραγματικά πρόκειται να δημιουργήσουν ένα νέο μέσο, μια νέα επιτροπή για την πολιτική συνοχής. Το είχαμε αυτό και πάντα τονούσε εκτός και αν θέλετε να δώσετε μια νέα κατεύθυνση, μια νέα όθηση. Αυτές λοιπόν οι δικές μου παρατηρήσεις και θα ήθελα να πω ότι η πολιτική συνοχής μας, η οποία μπαίνει σε μια καινούργια φάση, δεν μπορούμε να την καταδικάσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να εντείνουμε τις ε, σωστές αυτές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Να απαντήσει ο μιλητής. Um, uh, Αυτό που συνέβη κάποια στιγμή είναι συνηθισμένο στις πολιτικές. Δηλαδή τα κράτη-μέλη μάλλον δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τις πολύ θετικέ εμπειρίες κάποιων κοινοτικών πρωτοβουλειών που χρειάζονταν ένα mainstreaming. Και εκεί χάσαμε πολλά από τα, αυτά που είχαμε μάθει και ενδώσαμε στη γραφειοκρατία. Ίσως υπήρξε μια απόπειρα αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν μάλλον πιο πολιτική απόφαση. Και επίσης δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε το βαθμό κινητοποίησης ή ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων, ενώ προσπαθούσαμε να συγκεντρώσουμε τις πολιτικές αυτές σε λιγότερες προτεραιότητες. Και αυτό ήταν απαραίτητο, γιατί μιλούμε για ευρωπαϊκή πολιτική. Και αν δεν συγκεντρώσουμε μια κρίσιμη μάζα δημοσιονομικών πόρων και οικονομικών πόρων για ορισμένους τομείς, ο Ευρωπαίος πολίτης δεν θα δει τη διαφορά των πολιτικών μας γιατί η πολιτική μπορεί να συγχρηματοδοτεί καλά και κακά αποτελέσματα, αλλά ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, πώς θα συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που η ίδια δημιουργεί μερικές φορές. Και όταν είπα επιστροφή στις ρίζες, ενώ επιστροφή στη στιγμή εκείνη που υπήρχε mainstreaming των πρωτοβουλειών και που έγινε λάθος τον τρόπο που τις συμπεριλάβαμε στο mainstream. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα των μεταφορών. Για πολλές χώρες οι μεταφορές αποτελούν σημαντική ουσιώδη κοινοφελή υπηρεσία. Στην παρουσίαση της έκθεσης, οι μεταφορές εμφανίζονται ως δύο διαφορετικοί κλάδοι. Περιλαμβάνουν καταρχήν υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσουν το θέμα της καινοτομία, γιατί για να ευνοήσουμε την καινοτομία θα πρέπει να διευκολύνουμε τις συνδέσεις μεταξύ ενός βιομηχανικού κέντρου και ενός ερευνητικού κέντρου. Επίσης, επειδή υπάρχουν κάποιες θύλακες ηλικιωμένων, δεν μπορούμε να τους κρατούμε απομονωμένους, θα πρέπει και εκεί να βελτιώσουμε τις διασυνδέσεις. Μερικές φορές λοιπόν οι μεταφορές είναι μέσο για την επίτευξη άλλων γενικότερων στόχων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλα, όλα τα κονδύλια θα επικεντρωθούν στις βασικές προτεραιότητες, αλλά μόνο το 66%. Και κάθε χώρα θα είναι ε, ελεύθερη να αφιερώσει τους υπόλοιπους πόρους στους δικούς της στόχους και μάλιστα με πιο ελεύθερο τρόπο από ό,τι σήμερα. Υπάρχει υποχρέωση για τα δύο τρίτα των πόρων, αλλά το ένα τρίτο και η χρήση του ενός τρίτου απελευθερώνεται πλήρως. Σε ό,τι αφορά την εδαφική διάσταση. Η έκθεση έδειξε μετά από προσεκτική ανάγνωση της Πράσινης Βίβλου ότι η λέξη εδαφικός παίρνει τόσες διαφορετικές σημασίες γι' αυτό και αντί για εδαφική προσέγγιση, εδαφικό προσανατολισμό μίλησε για τοπικό προσανατολισμό, για τοπικό μοντέλο, place-based. Και έχετε δίκιο ότι η μονάδα αναφοράς της πολιτικής είναι μία περιφέρεια ε, με μικρό πι. Δηλαδή όχι μία περιφέρεια με τη διοικητική έννοια. Και δεν ξέρουμε τι στη περιφέρεια πριν ε, ξεκινήσει η εφαρμογή της πολιτικής. Γιατί ο καλύτερος τρόπος για να ορίσουμε μια περιφέρεια είναι ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο. Πρόγραμμα ίσον περιφέρεια. Ξεκινούμε ένα πρόγραμμα και από την αντίδραση που έχουμε από τους ενδιαφερόμενους, αν έχουν δείξει συμπληρωματικότητα, συνεργασία, ομοιογένεια, ομοιομορφία, τότε χάρη στο, με βάση αυτό το πρόγραμμα διαμορφώνεται και η ιδέα της περιοχής, της περιφέρειας. Το θέμα είναι γιατί μία έκθεση που αλλάζει τη μονάδα αναφοράς, ε, τι κάνει για τα ΝΑΤΣ 2 και για τον για την κατανομή των περιφερειών. Εκεί η έκθεσή μας ήταν πολύ συντηρητική. Γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε τα στατιστικά στοιχεία, ούτε την ε, κατανόηση, ούτε την πολιτική συνένεση για να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο τρόπο επιμερισμού των ε, κονδυλίων. Και αν ε, εμπλακούμε σε μια συζήτηση όπου θα προσπαθήσουμε να επινοήσουμε νέα μέτρα, θα καταλήξουμε σε μία φιλονικία μεταξύ των κρατών μελών και σε ένα διαγωνισμό ποιος θα απορροφήσει τα περισσότερα κονδύλια που θα είναι σχεδιασμένα με συγκεκριμένο ε, προγραμματισμό. Και η έκθεση λέει, από τη στιγμή που το κατόφλι του 75% είναι τόσο απότομο και πολλές φορές δημιουργεί κάποιους ε, στατιστικούς ελιγμούς, είπαμε να πούμε 75% συν χ, για να αποφευθεί αυτή η δραματοποίηση του 75%. Αλλά έχετε δίκιο, δεν είναι και πολύ συνεπές, αλλά αυτό γίνεται για πρακτικούς λόγους, γιατί η έκθεση προσπαθεί να μείνει προσγειωμένη και δεν προτείνει καμία αλλαγή του παρόντος επιμερισμού. Τώρα, για τον κανόνα των ταμείων προτείνουμε επαναφορά τους. Για, για το γεωργικό ταμείο, συγγνώμη. Για το ταμείο για την Ήπειθρο προτείνουμε επαναφορά του. Τώρα, για το κοινωνικό ταμείο προτείνουμε συγχώνευσή του με το περιφερειακό. Γιατί με τη μορφή αυτή και για ρεαλιστικούς λόγους λέμε ότι περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα λύσει μια συγχώνευση. Επίσης πολλά αναφέρουμε για τα χρήματα των φορολογουμένων στην έκθεση, γιατί μία από τη μορφή που ασκείται κατά της πολιτικής είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού χρησιμοποιούνται τα κονδύλια των φορολογουμένων. Γι' αυτό λέμε ότι τα τελευταία χρόνια παραδίνουμε έμφαση στον έλεγχο και την εποπτεία, που είναι σημαντικά θέματα, αλλά δεν μας λένε τίποτα για το πώς επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών μια συγκεκριμένη δράση και η χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου κονδυλίου. Ακόμη και τακτική δαπάνη κονδύλια να έχουμε, μπορεί παρόλα αυτά τα κονδύλια να μην εξυπηρετούν κάποιο σκοπό, να μην έχουν προστιθέμενη αξία. Εκεί επικεντρώνεται η έκθεση. Και δεν προτείνει. Δεν λέει ότι οι πολιτικές είναι αδιάφορες. Αλλά από ποιοτική άποψη, μερικές φορές δεν αντέχουν στις επικρίσεις. Για τις ορισμένους ε, τομείς, η ενίσχυση των ε, επιχειρήσεων και της καινοτομίας δείχνει ότι υπάρχουν αυτά αποτελέσματα. Τέτοιου είδους εκθέσεις θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα κονδύλια. Δηλαδή υπάρχει μελέτη των συνεπειών, των επιπτώσεων. Ξοδεύουμε κονδύλια για κάτι, να αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αυξήθηκε το δικαιωμένο προσωπικό, αυξήθηκε η, η, απασχολησιμότητα. Αυτό είναι, αυτά είναι απτά αποτελέσματα, να καταμετρηθούν. Όταν βέβαια λέμε ότι δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε ότι είναι δυσάρεστα τα αποτελέσματα, απλώς δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν αποτελέσματα. Οπότε δεν μπορούμε να δηλώσουμε ότι είναι αποτελεσματική η χρήση των κονδυλίων, των χρημάτων των φορολογουμένων. Και τέλος εκφράστηκαν ε, ανησυχίες για το θέμα που αντιμετωπίζονται οι αγορές από την έκθεση και το θέμα της απασχολησιμότητας και των επιχειρήσεων. Η έκθεση προτείνει την απελευθέρωση των αγορών ως σημαντικό στοιχείο της ειρήνης και της ευημερίας στην Ευρώπη. Και επιστρέφοντας στις ρίζες, διαπιστώνουμε ότι για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να συνεπικουρηθεί από μια αναπτυξιακή πολιτική. Το βλέπουμε αυτό στις αγορές οι αγορές ε, υφίστανται τέτοιες ε, πιέσεις σε ορισμένες περιφέρειες που δεν μπορούν να να χρησιμοποιώντας τη γνώση τους και εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογίες. Γιατί πολλές φορές είναι αντιδραστικές στην αλλαγή αγορές και ασκούνται πιέσεις ε, για να φημωθεί η απελευθέρωση των αγορών, να πληγεί στα σπάργανα. Αυτή είναι η παλιά ιστορία. Αλλά αν υπάρχει αναπτυξιακή πολιτική που θα συνεπικουρεί μια απελευθέρωση των αγορών, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πόροι για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Και μάλιστα υπάρχει ένα κεφάλαιο και ένα πολύ σημαντικό έγγραφο και για την καινοτομία. Η Ευρώπη, κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη της έκθεσης, δεν κατάφερε να υιοθετήσει μια συγκροτημένη πολιτική καινοτομιών και έρευνα. Έχει τα προγράμματα καινοτομία και έχει και τα ερευνητικά προγράμματα, αλλά δεν υπάρχει μια ενιολογική σύνδεση μεταξύ του. Θα πρέπει να βρεθεί ένα καλύτερο τρόπο για να συνδεθεί το ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο, που στόχο έχει ε, του πόλου αριστεί με τα προγράμματα των καινοτόμων περιφερειών, που έχουν στόχο την προσαρμογή της τοπικής γνώσης, της καλύτερης τεχνολογίας, της βέλτιστης τεχνολογίας και να αποφευθεί το λάθος κάθε περιφέρεια να ισχυρίζεται ότι έχει αριστεία, γιατί πολλές φορές έτσι εφαρμόζεται η πολιτική. Ο Γιάνν Όλμπριχτ. Κάποιος θα μπορούσε να συναγάγει το συμπέρασμα ότι θα πρέπει για να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι αδύνατο να τους υλοποιήσουμε. Ενδιαφέρον αυτό. Η έκθεση είναι ταυτόχρονα παραδοσιακή και πρωτότυπη. Θα σας ε, υποβάλω μια αφελή ερώτηση. Γιατί, αν κατάλαβα καλά, αν θέλουμε να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Αν θέλουμε μια εύρυθμη εσωτερική αγορά, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια αναπτυξιακή πολιτική. Αλλιώς δεν θα λειτουργεί εύρυθμη αγορά. Και η πολιτική συνοχή είναι απαραίτητη για τις αγορές. Κατά παράδοση και με βάση τη συνθήκη, για την εσωτερική αγορά μιλάω, ενιαία αγορά, την εσωτερική αγορά. Στην ε, ε, συνθήκη όμως κατοχυρώνει την πολιτική συνοχή ω πολιτική για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και των ισορροπιών. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τμήμα τη πολιτικής συνοχής ή της κοινωνικής συνοχής. Αλλά όταν λέμε στη συνθήκη μείωση των ανισοτήτων, εννοούμε μείωση των ανισοτήτων που δημιουργούν κολλήματα στην εύρυθμη εσωτερική αγορά. Ενώ για εσά η αναπτυξιακή πολιτική είναι αυτή που μειώνει τις ανισότητε και άρα έρει τα εμπόδια στην αγορά. Α, δεν έχουν όμως την ίδια γνώμη όλοι οι πολιτικοί ότι η μείωση των ανισοτήτων ισοδυναμεί με αναπτυξιακή πολιτική. Θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη εξήγηση και διευκρίνηση, γιατί μη θα επανέλθουμε στην παλιά συζήτηση για τις θεωρίες της περιφερειακής πολιτικής, για το ποιοι είναι κινητήριοι μοχλοί και ποιοι είναι οι πιο μειονεκτικοί. Αλλά εσείς θέλετε να αποφύγετε αυτή την παραδοσιακή αντιπαράθεση. Δεύτερον, η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί κατάλαβα καλά, εμείς μιλούμε πάντα για οριζόντια πολιτική συνοχής και εσείς προτείνετε πολυτομεακή πολιτική. Δεν είναι μόνο σημειολογική διαφορά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους μεγάλες τομεακές πολιτικές με καλές, καλά καθορισμένες τρεις-τέσσερις προτεραιότητες και αυτές οι προτεραιότητες θα εφαρμόζονται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες, όχι πάντα το ΜΕΚΕΣ. Αυτό το τμήμα θα έχει τοπικό προσανατολισμό, όχι γεωγραφικό. Γιατί πολλές φορές μιλούμε για εδαφική συνοχή. Τοπικό προσανατολισμό μιλούμε με τον κόσμο, σε συνεργασία με τον κόσμο. Γιατί δεν είναι όλα τομεακά. Έχουμε τομεακά αφενό και πολυτομεακά αφετέρου. Και μπορεί να έχουμε πολυτομεακά με τη συνεργασία του κόσμου. Γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ούτε την αναπτυξιακή πολιτική, ούτε να μειώσουμε τι ανισότητε. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Εκεί υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσε προτάσει. και ίσω και φιλοσοφία ολόκληρη, όχι μόνο λόγια. Λέμε πολυτομεακό ταμείο, ταμείο στον ελληνικό. Ένα μόνο ταμείο με τοπικό μοντέλο, πολυτομεακό ταμείο και τοπικό μοντέλο. Είναι παραστατική αυτή η πρόταση για ένα ενιαίο ταμείο. Ναι, όντως, αν θέλουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα, θέλουμε ένα ενιαίο ταμείο για πολυτομεακό μοντέλο. Αυτό όμως θα εξοργήσει πολλούς, φαντάζομαι. Αλλά είναι πολύ σημαντική η πρόταση. Κάτι άλλο που ίσως είναι μόνο συντακτικό, αλλά μπορεί και όχι, αφορά τις συμβάσεις ή την ε, πολιτική των συμβάσεων και επιχειρησιακά προγράμματα που θα εμπλέκουν τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τις περιφέρειες. Τι σημαίνει τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τις περιφέρειες. Δηλαδή θα είναι συμβάσεις με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Και το mainstreaming, πού το βάζετε. Είναι μόνο φραστική διατύπωση ή μιλάτε για διαφορετικές συμβάσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών ή και συμβάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις περιφέρειες τα... Ή μήπω θα είναι συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη και μέσα αυτών των συμβάσεων θα καλύπτονται και οι περιφέρειες. Μπορεί να είναι αφελείς οι ερωτήσεις μου, αλλά δεν ξέρω, είναι μόνο φραστικές αυτές οι, οι διατυπώσεις ή κρύβουν και μια φιλοσοφία. Ο κύριος Βανίστερ Ρόι. Νομίζω ότι τα σημαντικά θέματα που με απασχολούν, τι να σε κάποιες περιπτώσεις, σε, από κάποιες απόψεις ε, αποτελεί μια επιστροφή στα θεμελιώδη. Αλλά μήπως αυτό θα μπορούσε να γίνει με τα μισά κονδύλια, λύνουμε έτσι τα προβλήματα του μέλλοντος. Ή μήπως υπάρχει κάποια σχέση. Αν δεν ε, χρησιμοποιηθούν πλέον κονδύλια για τις υποδομές, μην μου λέτε ότι χρησιμοποιείτε κονδύλια για τα παιδιά, μιλάμε για ευημερία. Τον πυρήνα της ευημερία. Τι είπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υποβάλλατε την έκθεσή σας. Γιατί αυτοί σας ε, πλήρωσαν για την έρευνα αυτή. Τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον, λοιπόν. Πήρατε απάντηση. Ποια είναι η επίσημη, ο επίσημος χαρακτηρισμός της έκθεσης αυτής και για την Επιτροπή μας δηλαδή, γιατί θέλουμε να ξέρουμε ε, την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι... Αν ενισχύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πληρώνει 100% αν είναι πάρα πολύ ισχυρή, αν ε, κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση. Άραγε, 90%. 80%. Αυτό το ερώτημα να ανακύπτει, θεωρώ. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Και ότι είναι έκθεση στο Κοινοβούλιο για την ε, περιφερειακή συνοχή. Εσείς λέτε place-based. Καλό, καλό ιδέα. Αλλά ποιες είναι οι αρχές πίσω από την ιδέα αυτή, γιατί δεν μπορούν όλοι να προβούν σε τέτοιες δραστηριότητε. Αν θέλουμε να υπάρχει μία σχέση με την υπόλοιπη Ένωση, με τις ε, πιο πλούσιες περιοχές. Κρατάτε πολλά στοιχεία για το εθνικό εισόδημα, για παράδειγμα, αλλά για το στόχο 2 και 1 το κρατάτε αυτό ή προτιμάτε να εξαφανιστεί πρόεδρος την ε, Μποστινάρου, τελευταίο στον κατάλογό μας. Αν υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο, παρακαλώ να μας το πείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μπάρκα. Θα περάσω στα ρουμανικά, για να έχω μιλήσει συνολικά τρεις γλώσσες. Η πρότασή σας, η πρότασή σας για μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής φαίνεται να είναι η αρχή μιας συνολικής συζήτησης για το προφίλ γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς θα ξεφύγει και από την οικονομική κρίση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα με την πολιτική ανάπτυξη και με βάση το τι συμβαίνει στο διεθνές προσκήνιο με την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι αναπτυξιακέ του πολιτικέ που βασίζονται στι υποδομέ, στην προστασία του περιβάλλοντο, στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη. Βλέπουμε πως όλα αυτά συνδυάζονται. Οι πολιτικές λοιπόν αυτές, οι αναπτυξιακές της Κίνας και των ΗΠΑ τους επιτρέπουν να έχουν πιο χειροπιαστές απαντήσεις που σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εξαρτάται από τις αποφάσεις του εθνικού επίπεδου. Έπειτα, καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι σημαίνει, Σημαίνει ολοκληρωμένη προσέγγιση και συνεπή προσέγγιση συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου της Ανάπτυξης της ε, το οποίο θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο μέτρων. Και όπω ε, και ο συνάδελφό μα, ο Ζαν Μποπουή, ο οποίο είναι και συντάκτη μια άριστη έκθεση, η πολλαπλή διακυβέρνηση και οι πολλαπλέ εταιρικέ σχέσει είναι μια διέξοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον είναι πιο ισχυρή, θα πρέπει να είναι εκείνη το εργαλείο που θα φέρνει πέρα σε αυτή την πολιτική. Αυτό μας λέτε. Επίσης, ε, το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που θα αποσπάσουμε από την διαδικασία διαπραγματεύσεων, διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει από το Γενάρη του 2009 και θα ολοκληρωθούν στο τέλος της φετινής χρονιάς. Διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτικών κομμάτων του Κοινοβουλίου. Πού θα οδηγήσουν όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα έχει προκύψει, η νέα Επιτροπή, στα τέλη της χρονιάς, συγκεντρώνει όλες τις συνθήκες για να είναι τόσο ιδανική όσο, όσο τη θέλετε. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένο εάν στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων η ευρωπαϊκή διάσταση έπαιρνε μεγαλύτερη σημασία και η εθνική λιγότερη. Κύριε καθηγητά, να σας πω ότι του χρόνου θα συζητήσουμε για την αναθεώρηση, την ενδιάμεση αναθεώρηση και τις νέες τάσεις για το μέλλον το κοινοβούλιο μα θα πρέπει να εγκρίνει μια νέα πολιτική συνοχής για το διάστημα μετά το 2013. Πάλι θα ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Θα υπάρχει ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πολιετές, νέος στρατηγικός προγραμματισμός, νέος προπολογισμό, νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ εθνικών αρχών και ευρωπαϊκών και νέα εμπόδια. Πώς θα συμφιλιώσουμε εδώ τόσα διαφορετικά συμφέροντα τα συμφέροντα εννοώ των παλαιών και των νέων κατών μελών. Σε αυτό μάλιστα το νέο πλαίσιο, όπου το χάσμα συνεχώς βαθαίνει εξαιτία και τη οικονομική κρίση. Χαιρετίζω λοιπόν τη σημερινή σα ε, παρουσίαση και ελπίζω ότι βάσει αυτή τη μελέτη θα προοδεύσουμε ώστε να βρούμε μία λύση σκόπιμη για την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπάρκα. Ευχαριστώ. Ναι. Ένα από τα μείζωνα ζητήματα που έχουν τεθεί επιτάπητο είναι ποια είναι η βασική επίθεση κατά τη πολιτική αυτή, το βασικό επικριτικό σχόλιο. Ένα τρίτο τη παγκόσμια τράπεζα, και το λέω αυτό γιατί στην παγκόσμια τράπεζα υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ απόψει. Ένα τρίτο λοιπόν των μελών τη παγκόσμια τράπεζα υπέβαλαν μια έκθεση γεωγραφική, η οποία λέει ότι κάθε πολιτική πρέπει να έχει στόχο συγκεκριμένους χώρους, τόπους και συγκεκριμένες αγορές. Γιατί, γιατί όπως και η δική σας παραπομπή μας είπε, καταλήγουμε να δημιουργούμε ή μάλλον να παρεμποδίζουμε την ελεύθερη ροή κεφαλαίων και δυναμικού από περιοχές που δεν έχουν ε, μεγάλη επιτυχία προς τα αστικά κέντρα. Αυτό είναι και ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο η έκθεση προτείνει και υποστηρίζει ότι θα ήταν μεγάλο σφάλμα για όλη την περιφερειακή πολιτική να έχουμε στόχο μόνο τη σύγκληση. Η σύγκληση δυστυχώς είναι η έκφραση που έχει χρησιμοποιηθεί ως τώρα χρησιμοποιείται στη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Η σύγκληση ή το κατακεφαλή εισόδημα των περιφερειών δεν θα πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι ο στόχος αυτής της πολιτικής. Είναι απόλυτα σαφές. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό λέει η έκθεση. Γιατί? Γιατί στόχος των πολιτικών αυτών, όπως και η συνθήκη μας ε, δείχνει το δρόμο, και τι κάνουν και οι Αμερικανοί με το Σύνταγμά του. Α του κοιτάξουμε. Το ερμηνεύουν. Περνάνε αρκετό χρόνο στην ερμηνεία του. Η συνθήκη λοιπόν λέει ότι η πολιτική συνοχή πρέπει να στοχεύει στην ερμονική ανάπτυξη και την ε, άμπλυνση των ανισοτήτων. Τι σημαίνει ανισότητε. Ε, επί τη ουσία ευκαιρίε που έχουν οι πολίτε για να αντιμετωπίσουν τι αλλαγέ. Εάν οι ευκαιρίε προ του πολίτε δεν είναι παρόμοιε, τότε η όλη ένωση δεν λειτουργεί. Η αγορά δεν λειτουργεί εύρυθμα. Τίποτε άλλο δεν λειτουργεί. Οι πολίτε τη Ευρώπη αυτό περιμένουν από την Ευρώπη. Όχι να είναι ίσοι, αλλά να έχουν ίσες ευκαιρίε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τι σημαίνει να έχουμε ίσε ευκαιρίε, Ότι οι πολίτε άσχετα από το που κατοικούν στην Ευρώπη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν... Δύο πράγματα. Εάν οι περιοχή τους πληγεί από ένα πρόβλημα, μια κρίση, επειδή είναι φτωχή, επειδή είναι πλούσια, τότε θα υπάρξουν αυτομάτως εργαλεία που θα τις επιτρέψουν να υπερπηδήσει το εμπόδιο. Αυτό είναι αποδοτικότητα, αυτό είναι ανταγωνιστικότητα, να υπάρχουν συγκριτικά πλέον εκτήματα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η ισότητα. Ότι, να ξέρουν όλοι ότι θα γίνει προσπάθεια στις Βρυξέλλες, ώστε οι συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικά υποφερτές συνθήκες διαβίωσης, είναι κάτι που επιδιώκεται. Αυτό πολύ σωστά μέσω της μέθοδου, μεθόδου συντονισμού έχει επαναληφθεί και έχει καταδειχθεί με σαφήνεια. Τι άλλο αναφέρει ο πρόεδρος Μπαρόζ όταν μιλάει για τις προτεραιότητες του, για την ατζέντα του και με αφορμή τη νέα του εκλογή. Ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να ασκούν τα δικαίωμά τους. Ο Τόνι Άτκινς, θυμηθείτε, είναι πολύ λαμπρότερο η προσωπικότητα από ότι εγώ ίδιος. Θυμηθείτε ότι είχε απαντήσει σε πολύ δύσκολα ερωτήματα. Ποια είναι τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Τι εννοούμε με αυτή την αναφορά. Ποιο είναι το όριο. Ο μέσος όρος εθνικών ή ευρωπαϊκών καθηκόντων και δικαιωμάτων. Και τα δύο είναι η απάντηση. Οι συνθήκε διαβίωση των εθνικών πολιτών έχουν πλέον ευρωπαϊκή διάσταση, διότι βρισκόμαστε σε μια υβριδική κατάσταση. Είμαστε και Ευρωπαίοι και εθνικοί πολίτε. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν οι πολίτε μάλλον πρέπει να γνωρίζουν κάτι για τα όρια αυτά. Υπάρχουν δύο ειδών ανισότητε που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και με συγχωρείτε που πήρα τέτοια παρακαμπτήρια εδώ, αλλά για να αντιμετωπίσουμε τι ανισότητε δεν είναι μόνο το θέμα να κοιτάξουμε τι διαφορέ στο ανακεφαλή εισόδημα. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για τη Σικελία λόγου χάρη και ότι το εισόδημα της Σικελίας συνεχώς μειώνεται. Και ότι το συγκρίνουμε αυτό με το Λονδίνο. Μα δεν συγκρίνονται τα δύο πράγματα. Το Λονδίνο μπορεί να μην λειτουργεί ω αστικό κέντρο και η Σικελία ω αστικό κέντρο ούτε και αυτή. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μόνο κατά κεφάλι εισοδήματα. Α υποθέσουμε ότι τα εισοδήματα αυτών των δύο περιοχών αυξάνονται, διότι και οι δύο τα πάνε πολύ καλά. Το Λονδίνο έχει πολύ καλέ επιδόσει. Η Σικελία επίση ξεπερνά τα εμπόδια τη, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό. Άρα το κατακεφαλή εισόδημα δεν είναι καλό δείκτη. Είναι άσχετο. Δεν είναι καλό δείκτη για να μετρήσουμε την ισότητα, διότι είναι μέσο όρο το κατακεφαλή εισόδημα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μια περιφέρεια πηγαίνει ποσοτικά έστω καλά και έχει ποσοτικέ επιδόσεις και ε, επανέρχεται η καμπύλη τη, μετά για ένα μεγάλο διάστημα σημαίνει ότι θα πάει πολύ χειρότερα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ο κοινωνικό αποκλεισμό αντιμετωπίζεται αν βελτιωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα. Είναι άσχετο το κατακεφαλή εισόδημα, λάθο η σύγκληση. Η πολιτική αυτή δεν είναι πολιτική κατά των αγορών, ωστόσο μπορεί να γίνει κάποιες φορές, αλλά δεν είναι, δεν είναι αυτός ο στόχος της. Σας ευχαριστώ λοιπόν που το τονίσατε το σημείο αυτό και με επιτρέψατε να επανέλθω. Είναι πολύ σημαντικό. Για το πολυτομεακό ταμείο. Δεν θα τα είχα πει καλύτερα από σας τον ίδιο. Προσυπογράφω πολύ στον τοποθέτησή σας. Εξαιρετική παρατήρηση. Και για τις προτάσεις και το πώς θα γίνει αυτό για το ταμείο, το ένα ταμείο, σας είπα, είναι δύσκολο να πει κανείς πώς θα υλοποιηθεί. Για τις συμβάσεις. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Διότι το χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση, συμβάσεις με τα κρατημέλη και τις περιφέρειες. Λοιπόν, είναι δύο ειδών οι συμβάσεις εδώ. Ένα, με τις ε, διαχειριστικές αρχές και άλλο με το σύνολο του κράτους μέλους. Με το στρατηγικό και εθνικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, στη σημερινή κατάσταση πραγμάτων, το Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα είναι, ένα, πολύ αδύναμο, είναι ισχνό, δεν είναι δεσμευτικό, είναι ένα πολύ ωραίο έγγραφο, αλλά δεν έχει συγκεκριμένου στόχου. Δεν είναι ισχυρό. Αυτό που προτείνει η έκθεση είναι να υπάρξουν δύο ειδών συμβάσει. Για κάθε κάτω μέλο, μία σύμβαση που να προσυπογράφει η Επιτροπή, το κάτω μέλο και σε πολλά κράτη-μέλη και ίδιε περιφέρειε επίση. Διότι πολλά είναι τα κράτη που έχουν ομοσπονδιακή οργάνωση, όπω η Ιταλία ή η Γερμανία. Προφανώ εκεί χρειάζεται και η υπογραφή των περιφερειών. Κάτι που ήδη έχει γίνει. Φέτο κιόλα. Σε άλλε χώρε όχι. Μπορεί τα πράγματα να είναι πιο διαδοχικά. Αλλά πρέπει να υπάρχει σύμβαση μεταξύ Επιτροπή και κράτου μέλου. Λειτουργικό πρόγραμμα σήμερα. Και πώ επιλύεται, πώ αντιμετωπίζεται ο κίνδυνο τη αντίφαση με την ταυτόχρονη σύναψη τη σύμβαση. Γιατί τώρα λέμε ότι όταν υπογραφεί το σχέδιο θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το πρόγραμμα. Όχι, πρέπει να λειτουργεί το πρόγραμμα ήδη και τότε να υπογράφεται η σύμβαση. Γι' αυτό θα είναι η σύμβαση αυτή, η σύμβαση σε επίπεδο κράτου μέλου και θα είναι και των διαχειριστικών αρχών. Με υπουργεία, οργανισμού και όλου του ενδιαφερόμενου φορεί. Μια διευκρίνηση. Δεν αμύφθηκα. Όχι γιατί δεν είναι γενναιόδορη η Επιτροπή, αλλά γιατί από δική μου πρωτοβουλία, από δική μου διάθεση, Ότι δεν με πλήρωσε κανεί ούτε η Επιτροπή, πλήρωσε το κόστος του ταξιδιού μου για να έρθω εδώ. Και το ξενοδοχείο που είναι απέναντι από το κτίριο της Κομισιόν. Αλλά όχι, με χρηματοδότησε το Υπουργείο Οικονομία και Οικονομικών της χώρας μου. Ξεκαθαρισμένο και αυτό λοιπόν. Για τι υποδομέ Χαίρομαι που το φύγετε διότι δεν θέλω να υπάρχουν εδώ παρενόησεις. Οι υποδομές είναι σημαντικότατη συνιστόσα των δημόσιων και κοινοφελών υπηρεσιών. Δεν μπορεί κάποιε φορέ ε, να παράσχει κανεί εκπαιδευτικέ υπηρεσίε χωρί αξιοπρεπή σχόλια, ούτε ε, μεταφορές, μετακίνηση χωρί μεταφορέ, ούτε καλέ συνθήκε διαβίωση, αν δεν επιφαντήσει κανεί τι περιφερειέ του. Κάτι που είδαμε πρόσφατα και στη Μεσίνη, λόγω χάρη. Ε, είναι λοιπόν απαραίτητη συνιστόσα οι υποδομέ, αλλά δεν είναι ο, αυτός καθεαυτό στόχο. Είναι ένα εργαλείο και μέσο πίσω από όλε τι προτεραιότητε τη έκθεση. Υπονοούνται υποδομέ ω θεμελιώδη συνιστόσα μαζί με τι μη υποδομές κιόλα. Όμως οι υποδομές είναι και πρέπει να παραμείνουν καθοριστική ενιστόσα. Δεν είναι μια κουβέντα που τη χρησιμοποιούμε έτσι, είναι ούτε ένα εργαλείο αυτός σκοπό. Δεν μετατοπίζουμε όμως, ούτε επινοούμε εδώ νέου στόχους ευημερία, ούτε αφηρημένου ούτε θεωρητικού Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι με την ετικέτα της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, που μπορεί κανείς να την ενισχύσει όσο θέλει και μετά με την ετικέτα της ε, ισότητας, περισσότεροι πολίτες θα μπορούν να ξεπεράσουν το όριο, το όριο της κοινωνικής αυτής αξιοπρέπειας, της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Πολλέ φορέ όμω για να το επιτύχει κανεί αυτό χρειάζονται σκληρότατε προσπάθειε και με κατάλληλη χρήση των υποδομών. Για στην σχετικά με την Επιτροπή. Όπως κάποιος θύμισε, ο ιστότοπος της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζο περιέχει όλο το σχετικό υλικό. Να σας προτρέψω να δείτε τα της ακρόασης, όπου και μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που πήραν μέρος, εξέφρασαν την έκπληξή τους για το πόσο αδύναμες είναι οι συνθήκες που θέτει, οι προποθέσει που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρξαν και κάποιε παρανοήσει κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, γιατί κάποια είναι λίγο δυσνόητα. Αλλά είπε το μέλο του IMF. Ουσιαστικά γράφεται λευκό επιταγέ και του απαντήσαμε ότι δεν είναι και τόσο πολύ εν λευκό, διότι υπάρχουν συγκεκριμένε και αυστηρέ διαδικασίε. Αλλά πραγματικά εκείνο εξεπλάγει μέχρι να καταλάβει πόσο δύσκολη είναι η Επιτροπή να πει όχι σε μια χώρα για το πώ θα χρησιμοποιήσει κονδύλια για μια συγκεκριμένη δράση προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όπω είπα προηγουμένω, επιμείναμε και εκεί πολύ να λέμε ότι αν μια χώρα δεν έχει ένα κατάλληλο σύστημα αξιολόγηση για την εκπαίδευση, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί κονδύλια για την εκπαίδευση. Τέρμα. Και αυτό σήμερα δεν συμβαίνει. Και αυτό απαντά και στη σχόλια των συμβατικών οικονομολόγων που μας λένε ότι οι πολιτικές μας έχουν ε, τα κατάλληλα πολιτικά εργαλεία και είναι φτιαγμένα για θεσμικά όργανα. Μα δεν είπε κανεί ότι εδώ τα θεσμικά όργανα δεν έχουν ρόλο να διαδραματίσουν. Αλλά δεν μπορεί κανεί να δημιουργήσει εκπαιδευτικό σύστημα αν δεν επικεντρωθεί στην πολιτική που θα στοχεύει στου τόπου. Στην τοποκεντρική πολιτική. Εδώ ένας όρος που δεν θα έπρεπε ποτέ να χρησιμοποιείται ίσω είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών. Μα είναι σωστό όρο αυτό, γιατί πάντοτε υπήρχαν ε, αντιστάσει κατά τη ε, διαφοροποίηση. Δεν μπορεί να λέει κανεί ότι αυτό θα ισχύει για μια χώρα που συμμετέχει εδώ και 10 χρόνια, για κάποιο άλλο, για κάποια άλλη. Όχι. Όχι, η διαφοροποίηση χρειάζεται. Αν ορισμού έχει ένα θεσμικό όργανο μια χώρα και άλλη δεν το έχει. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τις χώρες που ήδη έχουν σχεδιασμό, ήδη έχουν προγραμματισμό και έχουν ένα διαφορετικό σχέδιο, εάν έχουν περιφερειακό προγραμματισμό, ώστε να αξιοποιήσουν. Δυστυχώ, και το γνωρίζουμε, υπάρχουν μια σωρία εγγράφων περιττών που παράγονται. Και το ακούμε αυτό και από κάποιες πλουσιότερες περιφέρειες που κάναν το σχόλιο. Και τέλος, όχι, δεν προτείνουμε να αλλάξουμε τη σημερινή κατάσταση πραγματών. Ακόμα και αν αυτό ακούγεται πολύ ασυνεπές μου, είπα προηγουμένω. Το τελευταίο μου σχόλιο, το ακροτελεύτιο, είναι ότι η λογική της έκθεσης αυτής και η φιλοσοφία της Επιτροπής που μου ζήτησε να συντάξω την έκθεση αυτή ήταν και το πλαίσιο της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης, της αναθεώρησης του προπολογισμού. Για να δούμε αν τα κονδύλια χρησιμοποιούνται σωστά, αν δεν χρησιμοποιούνται, γιατί αν δεν αξιοποιήσουμε το διάστημα αυτό του επόμενου 7 μήνε, θα έχουμε διαπραγματεύσει περί κονδυλίων μόνο. Και αυτό είναι μια δυσάρεστη κατάσταση πάντοτε. Σα ευχαριστούμε πραγματικά θερμά. Δεν έχουμε ακόμα πολύ χρόνο στη διάθεσή μα και χρειαζόμαστε ακόμα 5 λεπτά. Να σα ευχαριστήσω. Να πω επίση εξ ονόματο των συναδέλφων μου ότι τον επόμενο χρόνο και τα επόμενα χρόνια ίσως θα συζητήσουμε τέτοια θέματα και οι θέσεις μας θα παρουσιαστούν και από την Επιτροπή. Θα κάνουμε και κανονικές ακροάσεις. Ήταν μία μήνυ ακρόαση αυτή μαζί σας. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας υποδεχτούμε εδώ για να ακούσουμε τα σχόλιά σας και τις θέσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αν θέλετε, μείνετε για δύο λεπτά ακόμα για να κλείσουμε την ε, συνεδρίαση. Να πάμε στο 14, στα διάφορα. Δεν έχω διάφορα. Να σας ανακοινώσω, δεν ξέρω αν θέλει κανείς να πάρει το λόγο για τα διάφορα, για το 15, για την επόμενη συνεδρίαση. 3 Νοεμβρίου το απόγευμα ξεκινάμε στις 3 και 4 Νοεμβρίου ξεκινάμε το πρωί. Ελπίζω λοιπόν να παρευρεθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις δύο αυτές ημέρες. Πέρα στη συνεδρία σας. Thank you very